έγινε μέλος της Επιτροπής στη θέση του κυρίου Παπακοσταντίνου. Οπότε όταν του δίνουμε το λόγο του κυρίου Παπακοσταντίνου δεν θα χάνουμε τόσο χρόνο, αλλά αστείο ήταν αυτό. Βλέπετε ότι είμαστε σε μεγαλύτερη αίθουσα σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτό το ίδρυμα να έχει κανείς μεγάλες αίθουσες στη διάθεσή του γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα με μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα αυτά που θα συζητήσουμε αύριο. Δεν μπορέσαμε δυστυχώς να αυξήσουμε τον αριθμό των γλωσσών ε, της γερμηνίας. Έχουμε πάντα 12 γλώσσες στη διάθεσή μας. Ξέρετε ότι στον τομέα αυτό της πολυγλωσσίας υπάρχει ένα συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς θα έλεγα για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Φαντάζομαι όμως ότι μπορεί να υπάρχουν μέλη απογοητευμένοι που δεν, απογοητευμένα μέλη που δεν βλέπουν τη γλώσσα τους στους ταλάμους διευμηνίας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση τη γλωσσική στο μέλλον. Περνάμε απευθεία στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων δηλαδή, με τον πρόεδρο της ΣΕΟΠΣ, τον Γκάμπριελ Μπερναντίνο. Είναι πρώτη φορά που έρχεται εδώ σαν πρόεδρος της ΣΕΟΠΣ αντικαθιστά τον Τόμα Στέφαν, πήρε μάλλον τη θέση του Τόμα Στέφαν με τον οποίο είχαμε καλές σχέσεις εργασίας στο παρελθόν και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω επίσημα τον Τόμας για όλες τις φορές που ήρθε εδώ, που πήρε το λόγο και για την γενεοδορία πνεύματος θα έλεγα την οποία επέδειξε στις παρουσιάσεις του. Και έχω κάθε λόγο να υποθέσω ότι το ίδιο ακριβώς πνεύμα συνεργασίας θα διέπει και τις παρεμβάσεις και την παρουσία συνολικότερα του κυρίου Μπερναντίνο. Θα πάρει το λόγο ο κύριος Μπερναντίνο για 10 με 15 λεπτά, θα κάνει την παρουσίασή του για το πού βρισκόμαστε σχετικά με το ΣΥΟΠΣ 2010 και τον ελεγκτικούς μηχανισμούς ή την ελεγκτική αν θέλετε αρχιτεκτονική και δίνω το λόγο αμέσως στον Γκάμπριελ Μπερναρντίνο. Γεια Είναι μεγάλη χαρά για μένα το να είμαι στο ναό της Δημοκρατίας στην Ευρώπη. Όπως είπε η Πρόεδρος, είμαι νέος Πρόεδρος της ΕΙΟΠΣ. Εξελέγει μόλις πριν ορισμένες εβδομάδες και ζητώ ταπεινά εκ των προτέρων συγγνώμη για τα λάθη που μπορεί να κάνω. Θα σας παρουσιάσω και κάποιες διαφάνειες κάποιες ιδέες που θα ήθελα να σας μεταφέρω για την Solvency 2, για το που βρισκόμαστε σήμερα, για την σημερινή κρίση και τα μαθήματα που παίρνουμε από αυτά, για το Solvency 2. Όπως γνωρίζετε, οι συστάσεις τις οποίες δίδουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούν τεχνικές ρυθμίσεις, ταξινομήσεις, εκλογιμότητα, κεφαλουχικές απαιτήσει ε, για τη φερεγγιότητα. Νομίζω ότι με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου έχουμε καταλήξει σε αρκετά θετικά συμβιβαστικά επίπεδα. Θέματα αμοιβών, στελεχών εννοείται, που είναι υποσυζήτηση τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία λοιπόν σχετικά με το Solvency 2, Φερεγγιώτης 2 αν θέλετε, τα οποία έχουν συζητηθεί. Το θέμα είναι η επεξεργασία των συστάσεων αυτών που προέρχονται από τις διαβουλεύσεις. Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά έγγραφα στη διάθεσή μας. Λάβαμε τουλάχιστον στη δεύτερη φάση άνω των 20.000 σχολείων. Τα συζητήσαμε αυτά και στις ομάδες εργασίας και στις ομάδες μελών του ΣΕΙΟΠΣ, ιδιαίτερα σε αυτήν της 29ης Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν αναθεωρήσει τις συστάσεις μας, έχουμε βελτιώσει τις συστάσεις αυτές, έχουμε λάβει υπόψη τις περισσότερες από τις συστάσεις τις οποίες λάβαμε μέσω των συνεισφορών σας Κάποια βασικά σχόλια που πρέπει να κάνω. Πρώτον, υπήρξαν κάποια σημεία θα έλεγα ανησυχίας σχετικά με τη συμβατότητα ε, του Solvency 2 με το προηγούμενο επίπεδο, το επίπεδο 1. Είναι υποχρεωτικό στις περιπτώσεις αυτές να υπάρχει μια κάποια ερμηνεία. Είναι τέτοιο το θέμα που το απαιτεί. Αυτό πήραμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάποια θέματα, ανεπίσημα 6-7 θέματα, όπου η ερμηνεία την οποία είχαμε κάνει ε, σε σχέση με το level 1, με το επίπεδο 1, δεν ήταν ακριβώς η ίδια με αυτήν την οποία δίδαμε στο Solvency 2. Ξεκαθαρίσαμε τέτοια επιμέρους θέματα, τα σκεφτήκαμε βαθύτερα αν θέλετε. Υπάρχουν, παραμένουν όμως ορισμένα προβλήματα θα έλεγα, στα οποία ίσως να χρειαστεί να επανέλθω αργότερα. Υπήρξαν ε, επίσης κάποιες θέσεις υπεραντίδρασης στην κρίση. Αυτό είναι προφανές ότι εμείς σαν ελεγκτές ε, προφανώς και λαμβάνουμε υπόψη μας το τι συμβαίνει με την παγκόσμια οικονομική κρίση. Υπήρξαν επίσης και κάποιες ανησυχίες για τη συμβατότητα την διατομεακή ε, και τις αιτιολογίες τις οποίες χρησιμοποιήσαμε εμείς ε, στις συστάσεις τις οποίες κάναμε. Το θέμα αυτό είναι αρκετά ευρύ και περίπλοκο και δεν αφορά μόνο το CRD. Αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει μια συμβατότητα ανάμεσα στις προτάσεις τις οποίες κάνουμε και η συμβατότητα αυτή θα πρέπει να χαρακτηρίζει το σύνολο των τομέων όπως και τον πιστοτικό σαν παράδειγμα. Και υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία είναι αμφισβητήσιμο το που ανήκουν, αν είναι πολιτικά θέματα ή τεχνικά θέματα ή τεχνοκρατικά αν θέλετε θέματα. Προφανώς εδώ έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ υψηλά ποσά, οπότε ακόμα και τα τεχνοκρατικά θέματα και ρυθμίσεις έχουν πολιτική σημασία. Αλλά είναι σαφές ότι η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε ήταν μια διαφανής διαδικασία και τελικά θα υπάρξει ένα κείμενο ανατροφοδότησης όλων των σχολείων τα οποία έχουν προηγηθεί. Ελπίζω να το δημοσιεύσουμε στο τέλος της εβδομάδας με όλες τις συστάσεις συμβουλές τις οποίες κάνουμε, εκθέτοντας όμως και την τεκμηρίωση που βρίσκεται πίσω από τις συστάσεις αυτές. Υπάρχει μια τρίτη σειρά συμβουλών, η οποία δημοσιεύθηκε στις 2 Νοεμβρίου για το Solvency 2, για το δεύτερο επίπεδο δηλαδή. Υπήρξαν κάποια θέματα σύγκριση στοιχείων ανάμεσα στο MCR και το SCR. Υπήρξαν επίσης ε, οι ομάδες οι οποίες ασχολήθηκαν με το δεύτερο πυλώνα και την απόσβεση των κραδασμών στον δεύτερο πυλώνα. Στο τέλος του χρόνου, πριν από το τέλος μάλλον του χρόνου, θα δούμε ακριβώς και το σύνολο των κριτηρίων που χρησιμοποιήσαμε. Τώρα για την κρίση. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση, είναι ένα δεγονός. Πρέπει να βγάλουμε όμως τα κατάλληλα συμπεράσματα. Το τι συμβαίνει στον τομέα των ασφαλιστικό τους τελευταίους μήνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια χειροτέρευση σε κάποιες θέσεις ε, της ε, σε σχέση με το Solvency 1, εν πάση περιπτώσει, με... υπάρχουν κάποιες μειώσεις σε θέσεις φερεγγιότητας, υπάρχει μείωση κερδών, μείωση και συγγνώμη κερδών, έχει υπάρξει επίσης και μείωση των περιουσιακών στοιχείων, αν θέλετε, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών οργανισμών, λόγω ακριβώς των προβλημάτων αυτών, σε επίπεδο έκθεση σε κινδύνους έχουν υπάρξει κάποιες σημαντικές εξελίξεις και λόγω ακριβώς της κρίσης στην οικονομία αυτό έχει αρχίσει να γίνεται αισθητό και στις ασφάλειες. Επίσης σε επίπεδο πάλι έκθεσης κινδύνων βλέπουμε ότι υπήρξαν κάποιες καταγγελίες συμβολέων συμβάσεων ασφαλιστικών. Αυτό είχε αρνητικές συνέπειες. Και ένα από τα θέματα είναι και τα χαμηλά ε, επιτόκια, το χαμηλό ύψος των επιτοκίων, επίπεδο επιτοκίων σήμερα. Αυτό είναι ένα προβληματικό ε, πεδίο λόγω ακριβώς ξέρετε κάποιων εγγυημένων αποδόσεων οι οποίες έχουν, ε, στις οποίες έχουμε δεσμευτεί, έχει δεσμευτεί η βιομηχανία. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο ασφαλιστικός τομέας και ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχουν διαφορετικά επιχειρηματικά πρότυπα, ακολουθούν διαφορετικά επιχειρηματικά πρότυπα και αυτό δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες. Ποια είναι τα μαθήματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε για το Solvency 2. Για... Ε, καταρχάς λέμε ότι χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα, ένα σύστημα το οποίο να εκτιμά σωστά τους κινδύνους, η αρχιτεκτονική την οποία χρησιμοποιούμε και στα πλαίσια της οποίας κινούμε θα είναι υγιής στη βάση της αλλά απαιτούνται κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις και βελτιώσεις. Προσπαθήσαμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε στη συστάση μας κάποια από τα μαθήματα της κρίσης αυτής. Καταρχάς έλεγχος, ενίσχυση ελέγχου και διακυβέρνησης, επιμένουμε σε αυτό, ενίσχυση ελέγχου και διακυβέρνησης αυτό είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε πλέον σοβαρά υπόψη. Συνολική, ολιστική αντιμετώπιση ε, στους κινδύνους και στην έκθεση κινδύνους, σε κινδύνους. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο ε, κάποια συγκεκριμένα μέσα τα οποία έχουμε για να εκτιμούμε την κατάσταση, αλλά κυρίως να ε, μην αφήσουμε κανένα μέσο που είναι στη διάθεσή μας. Πρέπει επίσης να έχουμε περάσει και σε μια σωστή στάθμιση του SCR, Και τέλος πρέπει να διασφαλίσουμε μια εσωτερική δυναμική στα λεγόμενα εσωτερικά πρότυπα. Υπήρξε κριτική ιδιαίτερα στα χρηματοπιστωτικά συστήματα κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής Πρέπει λοιπόν το σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε να βασίζεται στα χρηστά πρότυπα των εσωτερικών αυτών διαδικασιών και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις δυνατότητες βελτίωσης των εσωτερικών προτύπων. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια μαθήματα τα οποία ξεπερνούν το Solvency 2. Τα προγράμματα σαν παράδειγμα εγγυήσεων στον τομέα των ασφαλιών. Είναι σαφές ότι τα προγράμματα αυτά σήμερα λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι πριν μερικά χρόνια. Η σωστή ενημέρωση των αυτών που υπογράφουν τα ασφαλιστικά συμβόλαια, των κατόχων των ασφαλιστικών συμβολέων, θα πρέπει να δίδουμε τη σωστή πληροφόρηση στους χρήστες και στους κατόχους και όχι να τους δίνουμε εκατοντάδες σελίδες ακατανόητες. Πρέπει να τους δίνουμε πληροφορίες οι οποίες να είναι κατανοητές, συγκρίσιμες και να τους επιτρέπουν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Σχετικά τώρα με τα κοινά έντυπα αναφοράς. Εμείς σαν Ευρωπαίοι ελεγκτές δεν έχουμε σωστές πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Ήταν πολύ δύσκολο να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία αυτά γιατί με διαφορετικό τρόπο συλλέγονται τα στοιχεία στις διάφορες χώρες. Και πρέπει να υπάρξει μια κάποια εναρμόνιση στα έγγραφα και έντυπα τα οποία χρησιμοποιούνται. Τέλος, κάποια από τα μαθήματα αφορούν και τον έλεγχο τον οποίο ανέφερα προηγουμένως αυτών των δραστηριοτήτων και σε επίπεδο βραχυπρόθεσμο και σε επίπεδο μακροπρόθεσμο. Τώρα εδώ βλέπουμε κάποια μαθήματα σχετικά με την έκθεση Λαροζιέρ και τους κανονισμούς της, την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι μπορεί να λειτουργήσουν θετικά. Είναι ο σωστός τρόπος συνέχισης της πορείας μας για τον έλεγχο της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού συστήματος αυτό θα οδηγήσει στην ενίσχυση και της νομισματικής σταθερότητας και της χρηματοπιστωτικής γενικότερα ηρεμίας. Δεν αφορά μόνο δηλαδή τις τράπεζες. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τις τράπεζες. Πρέπει να υπάρξει σωστή σύνδεση και αναλογία ανάμεσα στον έλεγχο ο οποίος θα γίνεται μακροοικονομικά αλλά και μικροοικονομικά. Θα πρέπει να συνδέονται οι δύο μορφές αυτές ελέγχου με τον σωστό τρόπο. Πρέπει να υπάρχει αναλογία στην ανταλογή πληροφοριών ανάμεσα στον μακροοικονομικό έλεγχο και τον μικροοικονομικό έλεγχο. Μετά, ε, ξέρετε ότι κάνουμε προτάσεις σε σχέση με αυτό το οποίο ονομάζουμε εγχειρίδιο κανόνων για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ενιαίο τέτοιο εγχειρίδιο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικές τεχνικές ρυθμίσεις, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές από τις αρμόδιες αρχές. Νομίζουμε δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα για τεχνικά επίπεδα ενιαία και δεσμευτικά, αλλά και για δυνατότητα βελτιώσεων από τις τεχνικές αρχές. Θέλουμε η διαδικασία αυτή συνολικά να οδηγεί ε, στην πλήρη δυνατότητα ελέγχου αυτών οι οποίοι λειτουργούν σε αυτόν τον τομέα, οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία, αλλά και να είναι πλήρως υπόλογοι έτσι ώστε οι ελεγκτές να μπορέσουν να λειτουργήσουν με τον σωστό τρόπο και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα από κοινού. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε υπόλογοι εδώ και απέναντί σας, απέναντι στο Κοινοβούλιο. Ένα ισχυρό μήνυμα από πλευρά μα είναι η ανάγκη για την εμπειρογνωμοσύνη η οποία προέρχεται από συγκεκριμένου τομεί. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα νούμερο για όλου, τα έλεγα Υπάρχουν πολλά επιμέρους στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και νομίζω η ιδέα την οποία ακολουθήσαμε για περισσότερες επιτροπές είναι η σωστή ιδέα για το μέλλον. και όταν μιλάμε για αρχές ελεγκτικές ευρωπαϊκές θα πρέπει να αποφύγουμε να φτιάξουμε αρχές πολύ μεγάλες, τόσο μεγάλες οι οποίες να γίνουν πλέον δυσδιαχείριστες. Ξέρετε ότι υπάρχουν δυνατότητες να ασχοληθούμε με διαφορετικό τρόπο με ορισμένα θέματα όπως τα πιστοτικά, όπως ε, τα χρηματιστηριακά, όπως τα ασφαλιστικά. Ξέρετε ότι ο ασφαλιστικός τομέας και η διαχείριση των ασφαλιστικών εισφορών είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι τελικά μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τομείς όπως το ασφαλιστικό και ε, για άλλους τομείς ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τομέα. Πρέπει να αποφύγουμε όμως τους πάρα πολύ μεγάλους οργανισμούς και επιτροπές. Τώρα για το πρόγραμμα εργασίας για το 2010. Ως συνήθως θα προχωρήσουμε την τεχνική μας δουλειά. Ταυτόχρονα επίσης θα προχωρήσουμε και στις αλλαγές τις οποίες έχουμε ξεκινήσει σχετικά με το Solvency 2 θα συνεχίσουμε. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια αυτή ελέγχου της φερεγγιότητας. Θα φτάσουμε στο τρίτο επίπεδο των διαπραγματεύσεων τον Φεβρουάριο του 2010. Αλλά ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μαζί, να σας ενημερώνουμε σωστά και εσάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο δεύτερο επίπεδο. Το είναι πάντα στη θέση που πρέπει έτσι ώστε να δίδει τις συστάσεις, συμβουλές και ιδέες οι οποίες απαιτούνται από πλευρά των πολιτικών εταίρων. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το QIS 5 Ξέρετε ότι αυτό το είχαμε συζητήσει και στα πλαίσια του Solvency 1. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τις συντάξεις θα δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν σε σχέση με αυτό σε πολιτικό επίπεδο. Εμείς περιμένουμε εδώ τις αποφάσεις του πολιτικού παράγοντα. Έχουμε επίσης μια ομάδα εργασίας η οποία θα δουλέψει καλά το 2010 για την προστασία του καταναλωτή. Έχουμε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για τη σύγκληση. Ξέρετε ότι και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι βασική προτεραιότητα για τον επόμενο χρόνο για μένα. Εφόσον πράγματι θέλουμε να εφαρμόσουμε σωστά το Solvency 2, το θέμα δεν είναι μόνο να γίνει γνωστό το θέμα αυτό και το πώς θα λειτουργήσει στους ασφαλιστές, αλλά και στους ίδιους τους ελεγκτές, στις ίδιες τις αρχές ελέγχου τις ίδιες τις ε, εποπτικές καλύτερα αρχές. Τότε μόνο η βοήθεια την οποία θα δίδει το ΣΕΙΟΠΣ θα είναι πράγματι χρήσιμη. Και στο τέλος η οικονομική σταθερότητα. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ανάλυσης της αγοράς, να δούμε από πού προέρχονται οι εντάσεις και να δώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες προς το πολιτικό επίπεδο και κατά τη διάρκεια του 2010. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα ήθελα σε μια πρώτη φάση να σας μεταφέρω. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και σχόλια. Σας ευχαριστούμε. Αν δεν σας πειράζει, θέλω να ακούσουμε πρώτον τον Πίτερ Σκίνερ, γιατί ήταν ο εισηγητής μας για τη Φερεγγιότητα 2. Και καλό θα ήταν να μιλήσει πρώτος. Είναι λογικό. Και σας προειδοποιώ ήδη ότι θα μιλήσει μετά η κυρία Περβάους Πέρες. Βλέπω ότι τα ίδια με το παρελθόν κάνουμε. Δεν έχουν αλλάξει συνήθειέ μα. Ευχαριστώ τον Καπριέλα Εμπονατίνη για την παρουσίαση. Τον συγχαίρω. Συγχαίρω και την Πρόεδρο. Για τα επόμενα βήματα επίσης θα είναι σκληρή η δουλειά μας και εργάζεστε σκληρά και είστε και δίκαιος, αυτό είναι γνωστό. Νομίζω ότι η ρεαλιστική σας προσέγγιση είναι η ιδανική για να εκπληρωθούν οι προσδοκίες μας σε σχέση με τον ΣΕΙΟΠΣ. Ελπίζουμε μελλοντικά ε, να λειτουργήσει αισίως ε, η, αυτή η εποπτική αρχή από το επίπεδο 1 όπου βασιζόμασταν στις αρχές όντως έχουμε παρεκκλίνει λίγο και πρέπει να καλύψουμε το κενό με συμβουλές τεχνικές που είναι απαραίτητες για διάφορους λόγους. Μας μιλήσατε για 20.000 απαντήσεις στη διαβούλευση. Εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα. Νόμιζα ότι ήταν 30.000 είναι δύσκολη η δουλειά σας και ελπίζω το επιτελείο σας να σε επικουρεί σε Αλλά υπάρχουν δύο ακόμη παράπονα ή μάλλον να το πω ζητήματα που σχετίζονται με τις ανακολουθίες που υπάρχουν και που ανέφερες και εσύ Γαμπριέλ. Για τη φερεγγιότητα 2 είπαμε ότι βασιζόμαστε στον κίνδυνο, αυτή είναι η προσέγγιση μας. Αλλά τι γίνεται με τις πτυχέ που βασίζονται στην ίδια την οικονομία, ποια είναι τα ωφέλη που αναμέναμε, οι οικονομικές μας φιλοδοξίες όταν εγκρίναμε την φερεγγιότητα 2 συνεχίζεται να επιδιώκεται τους ίδιους στόχους ή λόγω της τρέχουσας κρίσης ε, ε, θα έχετε αλλάξει πορεία. Βλέπω γνέφεται. Μιλώντας για τις ανακολουθίες και έχω και παραδείγματα να σας δώσω ένα συγκεκριμένο για το λειτουργικό κίνδυνο. Ε, για την ε, ε, αυξήσατε το κατόφλι από 30 σε 60% για τις κεφαλουχικές απαιτήσει. Αυτό όμως συνιστά ανακολουθία. Και τέτοια παραδείγματα και άλλα που θα προκύψουν κατά τη γνώμη σας σημαίνουν ότι επαναπροσδιορίζουμε τα κείμενα του επίπεδου 1 σε βαθμό που να πρέπει να αλλάξουμε και την φερεγγιότητα. Αυτό εξ αρχή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ε, δεύτερο σημείο τώρα που θέλω να σχολιάσω, η ίδια η οικονομική κρίση. Ε, χρειαζόμαστε μια συνεκτική προσέγγιση ε, για να καλύψουμε και τον τραπεζικό τομέα και τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Ε, και τι γίνεται σε αυτή η περίπτωση. Οι ασφάλειε παίζουν δεύτερο ρόλο έχουν υποβαθμιστεί σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό τομέα. Μήπω είναι υπερβολική αυτή η αντίδραση και πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία και να βρούμε για την κατάλληλη απάντηση. Για το ring fencing τώρα, για τι μη διασυνοριακέ συναλλαγέ, για χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά προϊόντα, κάτι που είχαμε συμφωνήσει στο επίπεδο 1. Θεωρούμε ότι είναι ένα περίπλοκο ζήτημα για τις χώρες και κυρίως για τις ασφαλιστικές εταιρείες που θέλουν να ακολουθήσουν, να αποδώσουν διαφορετική αξία στα στοιχεία του ενεργητικού τους. Ε, ε, πώς ακριβώς θα διαχειριστούμε αυτές τις περιπτώσεις, θα μπορούσατε να με ενημερώσετε και νομίζω ότι και εκεί χρειάζεται να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Τώρα, δύο ίσονο σημασία ζητήματα. Τι γίνεται με την αναλογικότητα, δεν έχουμε κανέναν ορισμό για τις μικρές εταιρείες ε, που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που πέφτουν κάτω από το κατόφλι της φερεγγιότητας διότι Τι θα κάνουμε με αυτές τις εταιρείες ε, και τέλος, χαίρομαι που ασχολήστηκε με τα καταναλωτικά ζητήματα. Καλό θα ήταν για τις ασφάλειες να υπήρχε υποπτική αρχή για τους καταναλωτές γιατί θα διευκόλυνε πολύ τη ζωή και το έργο μας. Ε, για την αντιστοιχία τώρα, την ισοδυναμία, την ambivalence ε, πρέπει κάπως να τοποθετηθείτε. Θα μπορούσατε να κάνετε κάποιες εισηγήσει. ή έστω να μοιραστείτε κάποιες ιδέες για να εξασφαλίσουμε την ισοδυναμία γιατί οι μιλάνε για ομοσπονδιακή αρχή, για τις ασφάλειες. Ε, πώς το σχολιάζετε παρακαλώ. Πίτερ, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Είναι σημαντικά τα ζητήματα και θα προσπαθήσω να εξηγήσω ποια είναι η θέση του ΣΕΙΟΠΣ για αυτά. Για το πρώτο σημείο, για την ανακολουθία σχέση με το επίπεδο 1. Αναγνωρίζουμε, όπως είπα, ότι σε κάποιους τομείς το κείμενο του επίπεδου 1 της φερεγγιότητας 2 μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό και γι' αυτό έχουμε διαφορετικά θεσμικά όργανα που εξετάζουν το κείμενο και προσπαθούν να βρουν τη σωστή ισορροπία. Σα διαβεβαιώ πάντως ότι για όλα τα ζήτημα που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου υποδεικνύει ότι αποκλίνουμε από το επίπεδο 1 Ε, προσπαθούμε να ε, εξετάσουμε και πάλι το κείμενο, να το δούμε από διαφορετική οπτική γωνία και ε, ορισμένες φορές αναγνωρίζουμε ότι είχαμε κάνει λάθος. Είχαμε βασιστεί για τον προσδιορισμό του κατοφλίου στους κινδύνους, στον κίνδυνο και στην ομάδα εργασίας αλλάξαμε γνώμη σε σχέση με αυτά που είχαμε προφασίσει στο επίπεδο 1 και έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα και συμπεριλαμβάνεται πλέον στις συμβουλές μας. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο όπου εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να αποδοθεί διαφορετική ερμηνεία σε σχέση με το επίπεδο 1. Πάντως λειτουργούμε πάσα διαφάνεια γιατί ακολουθήσαμε τις συμβουλές της Επιτροπής και για αυτά τα ζητήματα μέσα στο έγγραφο δεν έχουμε δώσει συμβουλές γιατί θα γίνει πολιτική συζήτηση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Οπότε για το καλό της συζήτησης είναι καλό να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ερμηνείες και σε πολιτικό επίπεδο θα επιλεχθεί το καταλληλότερο κείμενο για το επίπεδο 2. Ε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια πάντως για να μελετήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Για την χρηματοπιστωτική κρίση και τον αντίκτυπό της, ε, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η φερεγγιότητα 2 είναι αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά. Η προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το ισχύον σύστημα όπου δεν υπάρχει δυνατότητα αντιπαραβολής ε, ανάμεσα στα στοιχεία δύο χωρών γιατί είναι τόσο διαφορετικές οι προσεγγίσεις που ακολουθούνται. Ξακολουθούμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση του κινδύνου με αυτόν τον τρόπο ε, για ε, για την, τον ασφαλιστικό τομέα και για τους ασφαλισμένους τους ίδιους αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και ακριβώς τι έγινε με την κρίση. Αν το σύστημά μας βασίζεται στον κίνδυνο, πρέπει να δούμε τους κινδύνους της αγοράς. Δεν μπορεί να εθελοτυφλούμε και να μην, βλέπουμε, να μην αναγνωρίζουμε τι έγινε στην αγορά. Δείτε τι έγινε με τις κινητές αξίες και, τα, και την αντιστοίχηση ανάμεσα στα διάφορα ε, χρηματοπιστωτικά εργαλεία που υπάρχουν. Ξαναλέω, δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε και Φυσικά θα έπρεπε να παραπονιέστε αν δεν το κάναμε αυτό και αν δεν προσπαθούσαμε να εκδώσουμε ε, συμβουλές. Θα ε, προσπαθήσουμε να διέπεται το έργο μας από τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Δείτε τη διαβούλευση ε, για τα θέματα της calibration, της αντιστοίχησης. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλες, όλα τα τεκμήρια που είχαμε στη διάθεσή μας, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εποπτικές αρχές είναι, έχουν δίκιο για τα πάντα βασιζόμαστε στην ανάλυση και στα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και γνωμοδοτούμε. Αλλά φυσικά ε, προτιθέμεθα και θέλουμε να συζητήσουμε με τους διαφορούς ενδιαφερόμενους φορείς γιατί αν υπάρχουν άλλα στοιχεία για άλλου είδους κινδυνούς εμείς θέλουμε να γίνει διάλογος γιατί δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού. Τώρα αρχίζουν όλα αλλά φυσικά ε, δεν μπορούμε παρά να εξετάσουμε ακριβώς ε, πώς επλήγει η αγορά από την κρίση. Αυτό θα το κάνουμε. Για το ring fencing τώρα, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα για την προστασία των καταναλωτών και προσπαθήσαμε να συνεισφέρουμε. Υπάρχει ένα έγγραφο για το ring fencing και τις επιπτώσεις που έχει ε, αυτή η διαδικασία επί κάποιων στοιχείων της φερεγγιότητας 2 ε, προσπαθούμε να έχουμε τη σωστή προσέγγιση. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές ε, λύσεις και κάποια από όλες θα είναι η κατάλληλη. Για την αναλογικότητα θα θυμάστε ότι είναι, μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές το ζήτημα. Ε, στην ε, Πορτογαλική Προεδρία ε, παρακολουθούσα τη συζητή στο Συμβούλιο στην αρχή της Φερεγγιώτας 2 και το θέμα της αναλογικότητας θυμάμαι ότι ήταν ύψιστη προτεραιότητα και για το ΣΕΙΟΠΣ εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα. Μπορείτε να εφαρμόσετε την Φερεγγιώτα 2 με αναλογικό τρόπο και το ζήτημα για μένα ε, δεν είναι να ορίσουμε δύο συστήματα για τη φερεγγιότητα, 2, ένα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ένα για τις μικρές. Ε, δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα, είναι, θα είναι άδικο για τις μικρές επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές και ε, μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τη φερεγγιότητα 2 σε διάφορες επιχειρήσεις διαφόρων ειδών και έχουμε δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα πώς ακριβώς μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας τεχνικές διατάξεις. Μιλάμε για απλούστευση, για τον υπολογισμό των τεχνικών παραμέτρων, απλούστευση για τον υπολογισμό των κεφαλαιοχικών απαιτήσεων, για την ε, αποκάλυψη των στοιχείων, για την υποβολή αναφορών. Υπάρχουν στοιχεία που σχετίζονται με την αναλογικότητα και μετά την εφαρμογή ε, θα συνεχίσει να μας απασχολεί το ζήτημα, γιατί κατά τη γνώμη μου έτσι θα έπρεπε να υπάρχουν παραδείγματο χάρη στοιχεία από πλευρά των εποπτικών αρχών για τη νέα αρχιτεκτονική του συστήματο που θα συνιστούν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το πώς πρέπει να εφαρμοστούν τα επιμέρους ε, ε, τμήματα ε, τη φερεγγιότητα, διέχοντα κατά νου την αναλογικότητα. Για του καταναλωτέ, συμφωνώ μαζί σου, Πίτερ, είναι κρίμα και είναι ένα από τα ζητήματα όπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη δεν έχουμε καταφέρει αυτά που θα έπρεπε στο χρηματοπιστωτικό τομέα, διότι δεν έχουμε ένα πάνελ εκπροσώπων των καταναλωτών που να παρεμβαίνει άμεσα ε, και να ε, σχολιάζει και να κατακρίνει. Στο ΣΕΙΟΠΣ έχουμε ένα συμβουλευτικό πανέλ όπου υπάρχουν εκπρόσωποι των καταναλωτών ε, εκπονούν πολύ καλέ γνωμοδοτήσει και χαιρόμαστε που συμμετέχουν στι εργασίες του ΣΕΙΟΠΣ. Έχουν κρατέα θέση σε αυτό το συμβουλευτικό πάνελ, αλλά ε, ο, γενικότερα όταν εξετάζετε τέτοια συμβουλευτικά κείμενα, είτε προέρχονται από το ΣΕΙΟΠΣ είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δεν ε, θεωρώ ότι ε, έχουμε αρκετό feedback από τους καταναλωτές και πρέπει να το να ε, αναβαθμίσουμε την κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την ισοδυναμία θα εκπονηθεί έγγραφο. Τα κριτήρια για να κατοχυρωθεί η ισοδυναμία και ε, ευελπιστούμε να ε, είναι ε, καλό το έγγραφο για να κινηθεί η διαδικασία βάσει της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα. Από τεχνικής απόψης τώρα ασχολούμαστε με τα κριτήρια και νομίζουμε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ήταν μακροσκελής η απάντηση, αλλά πολλές ερωτήσεις σας. Η φαντάζομαι θα έχει και άλλες πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την εκλογή σας, το διορισμό σας για αυτό το θέμα που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και η νέα σας προσέγγιση σίγουρα θα είναι χρήσιμη. Ο Πίτερ Σκίνα που ήταν εισηγητής μας για τη Φεραγγιότητα 2, σας ρώτησε και απαντήσατε για το πώς ε, ερμηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επίπεδο 1. Όταν αποκλίνει, τη διορθώνεται. Εγώ θα περίμενα να πείτε ότι σε καμία περίπτωση ε, δεν αποκλίνεται από το επίπεδο 1. Απλώ θεωρείται το επίπεδο 2 ως τεχνικό στοιχείο. Και δεν ανατρέπεται ούτε διορθώνεται ο συμβιβασμός, ο πολιτικός συμβιβασμός που είναι στο επίπεδο 2 μέσω τεχνικών τροπών του επίπεδου 2. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση λιγότερο στον πρόεδρο του ΣΕΙΟΠΣ, αλλά στον κύριο ε, περισσότερο Γαμπρίελ Μπερναδίνο θέλω να κάνω την ερώτηση που έχει προσωπική άποψη και εμπειρία για ε, τα καθήκοντά του ε, ως ε, πρόεδρος του ΣΕΙΟΠΣ. Είπατε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πεδίο πέρα από τη φερεγγιότητα 2. Εγώ θα το χαρακτηρίζω ενδεχομένω και τα κατάλοιπα της φερεγγιότητας 2. Πώς θα το αντιμετωπίσετε άμεσα και επιγόντως σε σχέση με τα όσα γίνονται και σε άλλους τομείς, ας πούμε, ε, στις εγγυήσει των καταθέσεων. Δεν αρκεί απλώ να εξαγγέλουμε ότι θα γίνει αυτό. Παράλληλα, ε, πώς θα δράσετε πέρα από τι τράπεζε, υπάρχει ειδική ρύθμιση και ποια είναι αυτή κτλ. Δεύτερη ερώτηση, κάτι που δεν αναφέρατε, είναι το θέμα της ε, συζήτηση που θα ξανανοίξει γύρω από την οδηγία IOPR. Τι θα κάνετε και υπάρχει ανάγκη επίγουσα να ξανανοίξει αυτό το θέμα. Τρίτο θέμα, η ομάδα support. Τι γίνεται. Περιμένουμε να αναλάβουν οι εποπτικές αρχές, οι Λαροζιέρ ενω και ε, τότε από εκεί και πέρα θα αρχίσει η συζήτηση και αυτό θα είναι αρκετό ή μήπως θεωρείτε ότι είναι επίσης ε, το να περιμένουμε βλέποντας και κάνοντας το άλλο θέμα της ε, παρακράτησης. Φερακιότητα 2 όταν ήρθε δεν μας επέτρεψε να επιβάλλουμε στις ασφάλειες αυτά που είχαμε επιβάλει στις τράπεζες. Πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα και πώς θεωρείτε ότι μπορούν να μεταφερθούν αυτές οι διατάξεις και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Και ένα τελευταίο σχόλιο μου επιτρέπετε για την αναλογικότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ εδώ και να φροντίσουμε να συμβαστούμε αυτά που αποφασίστηκαν στο πρώτο επίπεδο. Γιατί εκεί ήταν όλη η συζήτηση. Δηλαδή, επειδή εγκρίθηκε η φερεγγιότητα 2, δεν σημαίνει ότι τώρα θα πρέπει να ασχοληθούμε ε, με την αγορά των μεγάλων τεσσάρων ή πέντε ανάλογα με το πώς ε, ε, αξιολογούμε τις εταιρείε, αλλά να υπάρχει και μια διαφοροποίηση και στην προσφορά και στην αγορά. Και μου φαίνεται περίεργο ότι η φεργιότητα 2 θα μας οδηγήσει σε υπερβολική ενασχόληση με τις ασφαλιστικές εταιρείε, ενώ συζητάμε και πρακτικά και θεωρητικά το πώς θα ε, αποφύγουμε το too big, too fair. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και σας. Έχω εμπλακεί πολύ σε αυτές τις συζητήσεις, ναι. Δεν είναι νέο ε, για μένα αυτό που βλέπω ότι οι ερωτήσει είναι πολύ ενδιαφέρουσες και εύστοχες και προκλητικές καμιά φορά. Για την, απόκληση, την παρέκκληση από το επίπεδο αναγνωρίζετε κυρία Μπερές ότι αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να αποστούμε από το επίπεδο 1. Το επίπεδο 1 είναι ένα κείμενο το οποίο όλοι έχουμε συμφωνήσει. Πώς να το πω. Και θα πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο λογικό. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ορισμένα θέματα όπου χρειάζεται ερμηνεία και το θέμα δεν είναι να επανερμηνεύουμε ή να ερμηνεύουμε με πολιτικό τρόπο κάποια θέματα. Υπάρχουν και τεχνικές συνέπειες και ορισμένα στοιχεία του κειμένου του επίπεδου 1 που χρειάζονται ερμηνεία όντως από πλευράς τεχνικών επιπτώσεων και μόνο. Και βεβαίως από πλευράς μας όπως σας είπα είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε με διαφάνεια και τη διαδικασία και βεβαίως μας ενδιαφέρει να παρέχουμε και συμβουλές έτσι, χρήσιμες στα ε, όρια βέβαια πάντα του επίπεδου 1 και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε ε, με παροχή συμβουλών το ε, πολιτικό πλέον επίπεδο να αποφασίσει. Εμεί δεν έχουμε καμία πρόθεση ούτε να ανατρέψουμε ούτε να αμφισβητήσουμε το κείμενο αυτό. Τώρα, για τα άλλα θέματα που αναφέρεται για τι εγγύησει των ασφαλιστικών ε, προγραμμάτων, σίγουρα υπολείπεται στην Ευρώπη ο κλάδος ο ασφαλιστικός σε σχέση με τον τραπεζικό, ας πούμε τι πιστεύει η ΣΕΙΟΠΣ Και αυτό το έχουμε πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την έχουμε συμβουλεύσει προ την κατεύθυνση αυτή, ότι χρειάζεται πηγόντω να αναλυφθεί η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, αν θέλετε, σταδιακή και βαθμία και να την παρακολουθείτε κι εσείς. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς να δούμε τι γίνεται στον τραπεζικό κλάδο. Για παράδειγμα, στις ασφάλειες ζωής. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις τράπεζες. Γιατί μιλάμε για προϊόντα που σε τελική ανάλυση είναι παρόμοια ε, με κάποια τραπεζικά. Λοιπόν, για τις ασφάλειες ζωής, αν τι άλλο, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη σύγκληση ε, με ε, τις λύσεις που έχουν δοθεί για τις τράπεζες. Ξέρω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα για το εάν και κατά πόσο θέλουμε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εγγυήσεων ή αν ε, όλα αυτά θα παραμένουν σε επίπεδο κρατών μελών. Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη η πολιτική απόφαση εδώ, αλλά τελικά κάποια στοιχειώδη σύγκληση θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων. Για τις υπόλοιπες ασφάλειες, εκτός από τις ασφαλείς ζωής, διαφέρουν τα πράγματα. Και εκεί βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει κάποια σύγκληση, αλλά είναι πολύ διαφορετική ε, αυτή ε, η ασφάλιση. Για τις ε, συντάξεις και τα ε, συνταξιωτικά ταμεία, pension funds. Και εδώ νομίζω εμείς ως Ευρωπαίοι χρειαζόμαστε, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση. Γιατί μου ζητήσατε να σας πω την προσωπική μου άποψη έτσι. Νομίζω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα σε μεγάλο βάθος. Τι θέλουμε να πετύχουμε τελικά αυτή η ιστορία των συντάξεων. Ξέρουμε ότι έχουμε πολλές διαφορές στα κράτη-μέλη, στις συντάξεις και στις ε, υποσχέσεις και τα δικαιώματα στην Ευρώπη. Όλοι θέλουμε εξασφαλισμένες συντάξεις, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε πού είναι η ασφάλεια αυτή. Υπάρχει πραγματογνωμοσύνη στα διάφορα εθνικά συστήματα, Έχουμε εργαστεί εμείς στο παρελθόν και για μας πολλές φορές είναι δύσκολο για τις ίδιες εποπτικές αρχές να κατανοήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν από χώρα σε χώρα στα συνταξιδοτικά συστήματα. Καλύτερα γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα συστήματα και είμαστε και πάλι πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Είναι πολύ σημαντικό ο τομέας αυτός για το μέλλον της Ευρώπης γιατί έχουμε και το δημογραφικό και τα λοιπά ε, θέματα, πρέπει να ασχοληθούμε. Τώρα, για τη φερεγγιότητα, υπάρχουν και άλλοι τομείς ξέρετε, που μπορούμε πολύ πιο εύκολα να ε, εργαστούμε για τις συντάξεις. Δηλαδή, παράδειγμα, πολλά από τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνου, αυτό που τώρα ονομάζεται φερεγγιότητα 2 για συστήματα διαχείρισης, διακυβέρνησης κτλ είναι κάτι που μπορούμε να μεταφέρουμε και να εφαρμόσουμε και στα αξιοδοτικά συστήματα. Γιατί όχι, σε μερικές χώρες ήδη εφαρμόζεται. Καλό θα ήταν αυτό και βελτίωση πιστεύω. Για την ομάδα support. Και αυτό θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε στο μέλλον. Και πάλι προσωπική μου άποψη είναι ότι όσο περνάει ο καιρό και όσο έχουμε μεγαλύτερη σύγκληση στα διάφορα συστήματα και η σύγκληση αυτή θα είναι καλύτερη με τα νέα εποπτικά συστήματα και τις νέες εποπτικές αρχές, αυτό το θέμα θα είναι πιο εύκολο, ελπίζω, στη συζήτηση. Ελπίζουμε στο προσεχές μέλλον. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι τα συστήματα εποπτείας εναρμονιστούν έτσι διαμιάς, ε, διαμαγείας. Δεν, δεν υπάρχει αυτό, δεν ισχύει, ας το παραδεχθούμε. Εγώ παρακολουθώ αυτά τα θέματα χρόνια ολόκληρα τώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θυμάμαι ε, από την αρχή τη συζήτηση έχει γίνει τεράστια, τεράστια σας διαβεβαιώ βελτίωση από τότε. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει και μεγαλύτερη βελτίωση και πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο μέλλον που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό στην ιδέα. Ε, για την αναλογικότητα τώρα. Τι να σας πω. Και στην εποπτεία σίγουρα οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει. Και ε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ένας τομέας από τον οποίο θα κριθεί η φερεγγιότητα 2 είναι πώς θα συγκλίνουν και οι εποπτικές αρχές στην Ευρώπη, διότι από το παρελθόν έχουμε αντλήσει και κάποια διδάγματα που λέγουν ότι μπορεί να είναι οδηγία ένα σύστημα στα χαρτιά και να αφορά όλη την Ευρώπη. Τελικά αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος που εφαρμόζεται η οδηγία αυτή. Είμαστε σε καλό δρόμο πιστεύω στη επιτροπή μας της ΕΙΟΠΣ για να καταλήξουμε τελικά σε ένα σύστημα εποπτείας ε, ουσιαστικά και γνήσια ευρωπαϊκό. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τη Φερογγιώτα 2. Και εκεί θα εφαρμόζεται και αναλογικότητα και βεβαίω χρειάζεται και στα συστήματα εποπτείας αναλογικότητα. Μας απασχολεί και στα έγγραφα που στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνουμε πολλές προτάσεις. Ένα τελευταίο τώρα για την εδραίωση, consolidation. Μήπω είναι υπερβολική η φερεγγιότητα δύο προς την κατεύθυνση ευθείας λύπης, όχι. Εγώ που παρακολουθώ αυτό το θέμα από την αρχή πιστεύω ότι θα υπάρξει και χώρος για διαφορετικές εταιρείε για διαφορετικούς ε, φορεί. και Η ε, εφαρμογή θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Ε, δεν σημαίνει ότι θα οδηγήσει απαραίτητα σε ενοποίηση εταιριών. Ας δούμε πώς θα ε, προχωρήσει στη πράξη και σε λίγα χρόνια νομίζω ότι ο κόσμος θα δέχεται περισσότερο έτσι με λιγότερη επιφύλαξη για την ιδέα αυτή. Αυτά. Thank you very much. Uh, next on my list is, is Udo. Ο Μπούλμαν. Μπούλμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Μπερναρτίνο, εγώ έχω δύο ερωτήσει. Πού, εν μέρη. Αν έχετε προβλήματα, να τα πω και αγγλικά. Όχι, όχι, όχι, όχι. Κανένα πρόβλημα, γερμανικά. Έχω δύο ερωτήσει. Εν μέρη ε, εν μέρη όχι. Συζητούμε εδώ για τις ασφάλειες τώρα, έτσι. Όχι μόνο για τις τράπεζες και για τις ασφαλιστικές εταιρείες στα πλαίσια της δημοσιονομικής κρίσης και για το πώς μπορεί κανείς να χαλιναγωγεί τους κινδύνους. Γιατί η νομοθεσία μας που συνεχίζεται και τρέχει θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σωστό πεδίο ε, για να ασκείται αυτή η δραστηριότητα, αλλά βλέπουμε πώς θα συγκρατούμε και τους κινδύνους. Το είπε και η κυρία Μπερές. Εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει η ευθύνη να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί πολλοί ενδιαφερόμενοι του κλάδου εμφανίζουν πολύ μεγάλες επιφυλάξεις αυτό. Ε, πολλοί φορείς λένε ότι εγώ αν είμαι πιο προσεκτικός από άλλους πρωταγωνιστές στην αγορά, γιατί να μοιραστώ τους κινδύνους με εκείνους που είναι πιο ρηψοκίνδυνοι και αναλαμβάνουν πολύ περισσότερους κινδύνους. Γιατί να, να φέρω εγώ την ευθύνη που έχω μια χρηστή διαχείριση και προσεκτική και έτσι έχω συνηθίσει να λειτουργώ στην αγορά. Αυτή είναι σημαντική ερώτηση, γιατί προχωρούμε προς μεγαλύτερη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια που είστε και εμπειρογνώμων, εσείς τι λέτε, ποια βήματα έχουν νόημα, ποια είναι άφρονα. Και μια δεύτερη ερώτηση, μια συζήτηση που γίνεται, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και αλλού, είναι κάτι που αφορά τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Πώς μπορούμε δηλαδή παγκοσμίω, μακροοικονομικά, να έχουμε συστήματα όπου εγκαίρως να εντοπίζουμε τους κινδύνους. τη στιγμή που γεννιούνται. Δηλαδή, ε, ένα συμβούλιο εκτίμηση κινδύνου, ένα risk board, λέγεται αυτό στα αγγλικά, που να εντοπίζει πολύ νωρί του κινδύνου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επιλέξει άλλο δρόμο. Λένε ότι υπάρχουν όργανα που ε, παρακολουθούν στη μακροοικονομική δραστηριότητα και τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιδοτικά ταμεία και όταν παράγουν πολύ μεγάλο κίνδυνο, το βλέπουν αυτό μακροοικονομικά. Εμείς τώρα έχουμε κάποιους οργανισμούς στην Ευρώπη. Πώς συνεργάζονται αυτοί για να εντοπίζουμε τους κινδύνους εγκαίρους και όχι κατόπιν εορτής. Πάρα πολύ αργά. Ευχαριστώ. Thank you um, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, ιδιαίτερα σχετικές με το θέμα που συζητάμε. Για την πρώτη, σχετικά με τα συστήματα εγγυήσεων στον τομέα των ασφαλιών. Έχουν ακουστεί πολλές κριτικές σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των συστημάτων εγγύησης και των προβλημάτων που μπορεί να διεφέρουν στην επιφάνεια αυτού του είδους τα συστήματα εγγύησεων ιδιαίτερα σε επίπεδο ασφαλιών ζωής. Τα συστήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα του σφαιρικού πλέον καθεστώτος. Και ο πιστοτικός τομέας και ο ασφαλιστικός τομέας και ο επενδυτικός τομέας εν πολλής ανταγωνίζονται ένα ένας τον άλλον στο ίδιο τμήμα της αγοράς. Αναζητούν η ίδια κεφάλαια, τις ίδιες επενδυτικές δυνατότητες και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ή εν πάση περιπτώσει να είναι συμφατά τα επίπεδα προστασίας αυτής της δραστηριότητας και των επενδυτικών ταμείων και των ε, πιστοτικών οργανισμών και των ασφαλιστικών εταιριών. Το θέμα λοιπόν είναι σε μια πρώτη φάση να υπάρχει η κατάλληλη αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας των καταναλωτών για όλα τα είδη των προϊόντων αυτών. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά και πώς θα συνδυαστούν τα διαφορετικά στοιχεία τα οποία συναποτελούν αυτά τα προγράμματα εγγύησης, τα σχήματα εγγύησης. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς πολλά μέσα, το μέσο της χρηματοδότησης, το μέσο της διόρθωσης και απαλλαγής από ορισμένα αντικίνητρα τα οποία υπάρχουν. Υπενθυμίζω ότι σε ορισμένες χώρες αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται σε αναλογικό επίπεδο αντιθέτως του κινδύνου το οποίο προκαλούν στο σύστημα. Ενώ θα πρέπει ε, να γίνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τους κινδύνους τους οποίους εκτίθεται το σύστημα και είναι πλέον σαφές ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα επιμέρους θετικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες για να καταλήξουμε στο κατάλληλο επίπεδο σύγκλησης των συστημάτων προστασίας του καταναλωτή στις δραστηριότητες αυτές στην Ευρώπη. Αυτό είναι κυρίαρχο θα έλεγα στην προσπάθειά μας. Η κρίση έδειξε ότι σε ορισμένες χώρες οι αγορές και η βιομηχανία ήταν κατά ορισμένων μέτρων στο παρελθόν των κεφαλαιοχικών σαν παράδειγμα εγγυήσεων ε, κάποιων ε, επενδυτικών μορφών και συστημάτων και μέσων, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις τράπεζες σαν παράδειγμα. Τώρα για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και την μακροοικονομική ε, μορφή εποπτείας ή την μικροοικονομική μορφή εποπτείας. Αυτά είναι θέματα τα οποία καλύπτουν και τους τρεις τομείς, και τον πιστοτικό τομέα και τον ασφαλιστικό τομέα και τον επενδυτικό τομέα. Νομίζω ότι ο, ο μακροπρόθεσμος έλεγχος, ο μακροοικονομικός μάλλον έλεγχος είναι κάτι το οποίο απεδείχθη ότι είναι απαραίτητο πλέον. Προφανώς και θα πρέπει να έχουμε και τις απόψεις του πιστοτικού τομέα για την οικονομική σταθερότητα. Προφανώς και οι ασφάλειες όμως και τα συνταξιοδοτικά συστήματα όπως και οι θεσμικοί επενδυτές παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία του χρηματοπιστωτικού συστήματος μόνο και μόνο γιατί είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές στην Ευρώπη. Αν υποθέσουμε ότι θα αποεπενδύσουν τα κεφάλαιά τους τότε δεν θα μιλάμε για οικονομική σταθερότητα. Γι' αυτό παρακαλώ όταν αναζητείτε λύσεις σε σχέση με την μακροοικονομική μορφή ελέγχου και εποπτείας να μην ξεχνάτε τις ασφάλειες τον ασφαλιστικό τομέα και τον τομέα διαχείρισης των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. Η νέα εποπτική αρχή Ίσως να χρειάζεται περισσότερη, περισσότερη ενημέρωση θα έλεγα και περισσότερα στοιχεία εμπειρογνωμοσύνης από τον ασφαλιστικό τομέα. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο γενικά να μιλάμε για χρηματοπιστωτικούς κινδύνους, αλλά και για άλλες μορφές κινδύνου επιμέρους που δημιουργούν προβλήματα στην ισορροπία της αγοράς. Ένα σεισμός είναι ένας εξωγενής παράγοντας. Λοιπόν, απαιτείται να υπάρξει μια ισόρροπη λήψη υπόψη της εμπειρογνωμοσύνης του κάθε τομέα που μας απασχολεί σήμερα. Τώρα για την διασύνδεση και την αμοιβαία ενημέρωση της ε, μακροεποπτείας και της λεγόμενης μικρο ή χρονικά εποπτείας. Το θέμα είναι να παρέχεται η κατάλληλη ενημέρωση στην Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων για τις υπερβολικές εκθέσεις ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σαν παράδειγμα. Μία από τις μεγαλύτερες βελτιώσεις τις οποίες θα έχουμε είναι αυτός ακριβώς ο τομέας. Μέχρι τώρα στο ΣΕΙΟΠΣ δεν είχαμε την δυνατότητα να συγκεντρώνουμε σε μία τράπεζα δεδομένων όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε από πλευράς για το σύνολο της Ευρώπης, γιατί κάποιες χώρες μέλη και κάποια τμήματα του ΣΕΙΟΠΣ εθνικά δεν έχουν την δυνατότητα να μας δίνουν όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα όμως εδώ θα υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση. Θέλουμε λοιπόν τέτοιου είδους αποκεντρωμένες πληροφορίες, θέλουμε πληροφορίες οι οποίες να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και κατάλληλες για την ανάλυση που κάνει η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Απ' την άλλη το θέμα αυτό δεν συζητιέται πάρα πολύ, δηλαδή το θέμα της ενημέρωσης δεν είναι κάτι το οποίο α, συζητιέται πάρα πολύ θα έλεγα τον τελευταίο καιρό και ε, θα πρέπει η Επιτροπή αυτή να είναι σε θέση να ενημερώνει σωστά όλους τους εταίρους σε αυτή τη δραστηριότητα, όλους τους πρωταγωνιστές αυτής της δραστηριότητας. Μιλάμε λοιπόν για αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση. Ευχαριστώ. Επιτρέπω να μακρηγορούμε και σε επίπεδα ερωτήσεων και σε επίπεδο απαντήσεων γιατί έχουν μεγάλη σημασία όλα αυτά τα θέματα. Σιλβί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα απαντήσω στο αίτημά σας και θα εγκαταλείψω το ίμιση της ερωτήσεώς μου μιας και δόθηκαν ήδη κάποιες απαντήσεις στον κύριο Μπούλμαν. Είμαι η συγχύτρια για την Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου και ίσως θα μπορούσατε να μου δώσετε περισσότερες συγκεκριμένες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για θέματα τα οποία αφορούν τις ασφάλειες, αλλά έχουν κάποιες πιο ειδικέ θα έλεγα πλευρές όπως το θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τώρα, για το πόσο ε, έρχεται σε αντίθεση ή πώς μπορούμε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στον ενεξάρτητο χαρακτήρα των αναλύσεων αυτών και των εποπτικών αρχών οι οποίες τις επεξεργάζονται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ανεξέλεγκτες ε, μορφές λειτουργίας των επιτροπών αυτών που θα πρέπει να παραμένουν υπόλογες. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα σας δώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις σε εύθετο χρόνο για την πρώτη σας ερώτηση. Είμαστε ανοιχτοί πάντα στο διάλογο μαζί σας. Και θα υπάρξει η δυνατότητα στο μέλλον να σας κάνουμε συγκεκριμένες συστάσεις προτάσεις για το θέμα του υπολόγου και του ανεξάρτητου χαρακτήρα. Νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία έχει ήδη ε, δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι έχει συλλάβει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην υπευθυνότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει την αρχή αυτή και στην ανεξαρτησία της επίσης. Είπαμε ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε μια Ευρωπαϊκή Αρχή Ελέγχου ή Αποπτική Ευρωπαϊκή Αρχή, που να είναι πιο ανεξάρτητη αν θέλετε από το επίπεδο ανεξαρτησίας το οποίο ε, χαίρουν ε, τα μέλη της σε εθνικό επίπεδο. Προφανώς και η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να είναι υπόλογη και προς τις κυβερνήσεις και προς τα κοινοβούλια περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Επιτροπής ε, κάποια συγκεκριμένα χρήσιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες αυτές ασκούν τις δραστηριότητές τους. Θα πρέπει άλλωστε να επιβεβαιωθεί η θέση του Προέδρου αυτού της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο στο μέλλον. Όλα αυτά θα έλεγα διασφαλίζουν το υπόλογο της συγκεκριμένης ομάδας. Από την άλλη όμως θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την ανεξαρτησία της. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό πρέπει να βρεθεί μια κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συγκεκριμένων επιτροπών και του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στο εσωτερικό αυτής της Επιτροπής σε επίπεδο δεσμευτικών τεχνικών ρυθμίσεων σαν παράδειγμα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια σωστή ισορροπία και να αποφύγουμε κάτι το οποίο είναι τεχνικό από την ίδια του τη φύση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αγνοεί και να αλλάζει αυτές τις τεχνικές συστάσεις τις οποίες εμείς θα πρέπει να δώσουμε. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα λοιπόν επανεξέτασης για τη διασφάλιση της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στο τεχνικό κομμάτι και το πολιτικό κομμάτι. Έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ. Κάθριν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον για τη φερεγγιότητα 2 και τα περί ε, εισφορών ε, ρευστότητας, ε, liquidity premium. Αν δεν προβλεφθεί κάτι, θα ακολουθήσει κατ' εκτίμηση 20% μείωση που είναι εξαιρετικά επιζήμη για τους καταναλωτές και για τη βιομηχανία, για την προστασία των καταναλωτών. Πώς βλέπετε αυτές τις αδυναμίες σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και τι προτείνετε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα των ελλείψεων Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σας δώσω σύντομες απαντήσεις. Ε, εισφορές ρευστότητας, ναι, ε, σύντομη ερώτηση, αλλά μεγάλο θέμα. Είναι επιτάπητο στο θέμα και μάλιστα προέκυψε σε στο τελευταίο στάδιο των συζητήσεων αφού ε, είχαμε στείλει εμείς τις συμβουλές στη διαβούλευση συζητήθηκε το θέμα με τους εμπλεκόμενους φορείς για να δώσουμε τις πρώτες συμβουλές ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το έγγραφο που θα στείλουμε αυτή την εβδομάδα. Για το τεχνικό ζήτημα, αν ε, δηλαδή υπάρξει τέτοια εισφορά ρευστότητα, σε πού ακριβώς πρέπει να προβλεφθεί, είναι τεχνικό το ζήτημα. θα συζητήσουμε το θέμα, θα υπάρχει και task force για, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα δούμε αν ε, το επιτόκιο απελαγμένο από τον κίνδυνο θα επιβαρυνθεί με, αυτό, αυτή την εισφορά ρευστότητα και σε συνδυασμό και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα θα καταλήξουμε ως συνήθως στην κατάλληλη απόφαση γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αυτό το θέμα, γιατί είναι και τεχνικό και πολιτικό. Ε, γιατί το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλα πόσα όταν μιλάμε για τεχνικές διατάξεις. Θα δώσουμε τις συμβουλές μας πώς πρέπει να ενταχθεί αυτό το premium, δηλαδή στο γενικότερο σύστημα, αλλά τελικά πολιτική απόφαση θα ληφθεί. Εμείς θα συνεισφέρουμε με τις ε, γνώσεις μας και ελπίζουμε να συζητηθεί το θέμα με διαφάνεια. Θα μας απασχολήσει και έτσι θα εξελιχθεί η διαδικασία τους προσεχείς μήνες. Λοιπόν, η προστασία των καταναλωτών τώρα. Βλέπαμε τα σχόλια των καταναλωτών και τα εξετάσαμε γιατί έχουμε διαπιστώσει την έλλειψη της ισορροπίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει κάποια σχέδια, ούτω ώστε οι ομάδες να είναι πιο προσανατολισμένες στο το θέμα της προστασίας των καταναλωτών, ε, κυρίως επειδή είναι εξαιρετικά περίπλοκα τα ζήτημα. Είναι περίπλοκα τα ζητήματα από πλευρά ΣΕΙΟΠΣ. Αυτό που μας απασχολεί είναι οι διαφορετικές πραγματικότητες που ισχύουν στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πραγματική σύγκληση. Προσπαθούμε να αναλύσουμε την κατάσταση για να δώσουμε μελλοντικά συμβουλές. Θα μπορούσατε, λέει η Πρόεδρος, νωρίτερα να δηλώνετε ότι θέλετε να πάρετε το λόγο. Θα με διευκολύνετε πάρα πολύ. Ο Μία μικρή ερώτηση έχω, σύντομη μόνο. Αφορά τις μικρομεσαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Ε, την περασμένη εβδομάδα είχα πάει σε μια διασκεψία που συμμετείχαν και πολλοί υπάλληλοι τέτοιων μικρών ασφαλιστικών εταιριών και μεσαίων. Ρωτώ λοιπόν, Πώς θα βεβαιωθείτε όλες αυτές οι διατάξεις και συστάσεις ότι δεν θα επιβαρύνουν ιδιαίτερα αυτές τις μικρές και μικρομεσαίες ασφαλείς. Ο κόσμος ανησυχεί πολύ. Ευχαριστώ. Yes, thank you very Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Η απάντηση νομίζω είναι η αναλογικότητα. Το είπα και προηγουμένως. Αν δείτε στον όγκο των συμβουλών που δίνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε έγγραφο θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν αναφορές και συστάσεις για το πώς εφαρμόζεται η αναλογικότητα και στους τρεις πυλώνες, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και στην εποπτική διαδικασία. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η φερεγγιότητα 2 δεν είναι κάτι που μας απασχολεί μόνο από τη σκοπιά των μεγάλων εταιριών, των κολοσσών, όχι. Σε καμία περίπτωση και στην εφαρμογή θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε και όπως σας είπα χρειαζόμαστε πρακτικά ε, παραδείγματα για το πώς εφαρμόζεται η αναλογικότητα και αυτό τον καιρό συνεργαζόμαστε με τον κλάδο και με τις ενώσεις για να ε, έχουμε και τα στοιχεία. Είναι η διαδικασία ε, ανοιχτή και διαφανής, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα. Υποτίθεται ότι μου είχατε πει να μην κάνω καμία ερώτηση, αλλά χρειαζόμαστε τρεις τέτοιες αρχές. Δεν γίνεται με μία μόνο. Και η διευθέτηση διαφορών τώρα ανάμεσα στις εθνικές ε, εποπτικές αρχές. Ε, πώς θα χειριστείτε αυτό το ζήτημα και υποτίθεται ότι έπρεπε να αλλάξει ε, η προσέγγιση στην ε, Βρετανία, στην Ιταλία και στη Λιθουανία πρέπει να ισχύει η ίδια κουλτούρα, το ίδιο πνεύμα. Πώς ακριβώς θα το καταφέρετε αυτό. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις. Γιατί χρειαζόμαστε τρεις διαφορετικές αρχές. Στις διαφάνειες έβαλα κάποια επιχειρήματα για να σας εξηγήσω Υπάρχουν διάφορα ε, σημαντικά ζητήματα. Υπάρχει η τεχνογνωσία και οι ιδιαιτερότητες. Είναι αδύνατον κάποιο, κάποιοι να ασχολούνται με όλες τις ιδιαιτερότητες, όλους τους κινδύνους μέσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ε, γιατί είναι ε, πολλά και διαφορετικά τα προβλήματα και έχουν ε, διαφορετικές επιπτώσεις και υπάρχει και αλληλεπίδραση ανάμεσα σε, όλους, σε όλες τις οικονομικές παραμέτρους. Η ρευστότητα, το σημαντικότερο ζήτημα δεν έχει καμία σχέση με τον κίνδυνο ε, στις ασφάλειες όταν δεν μιλάμε για ασφάλειες ζωής. Εκεί υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ με άλλα τμήματα τη οικονομία. Χρειαζόμαστε πολλού και διαφορετικού ειδικού. Ναι, βέβαια μπορούμε να συνδυάσουμε του ρόλου του. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά τελικά θα έχουμε μια υπερφύαλη δομή που δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε. Οφείλουμε να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες βέβαια κάθε θεσμικού οργάνου και όταν γίνει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις επαγγελματικέ τάξεις και τις ασφάλειες ε, γιατί οι τράπεζες θα είναι σίγουρα στην κορυφή της λίστας αλλά τι θα γίνει μετά με τις συντάξεις και τις ασφάλειες. Αυτό είναι το θέμα. Για τη διευθέτηση των διαφορών τώρα θα είμαστε έτοιμοι πιστεύω αν ακολουθηθεί η δέουσα διαδικασία βέβαια και αυτό έχει σχέση με το έγγραφο που τώρα συζητείτε. Θα είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε το ζήτημα με επαγγελματικό τρόπο. Τώρα μιλήσατε για διαφορετική κουλτούρα και τα διαφορετικές ε, ε, προσεγγίσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, εντάξει νομίζω ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα με το έγγραφο, με τη φερεγγιότητα και το δεύτερο βήμα θα γίνει με τις εποπτικές αρχές. Ευχαριστούμε. Μόνο εγώ υπολείπομαι στον κατάλογο ε, των ομιλητών. Ε, με πρόλαβαν οι συνάδελφοι, αλλά θα ήθελα ε, να σχολιάσω κάποια, κάποιες από τις απαντήσεις σας το ότι θα έχουμε τρεις διαφορετικούς οργανισμούς και ε, εξετάζοντας και το ιστορικό υπόβαθρο της ε, θέσπισης τους ε, κατάλαβα ότι μας είπατε πως παρα, παραγωνίζεται συνήθως ο ασφαλιστικό τομέας σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα. Και όπως είπατε, οι ασφάλειες είναι και ο μεγαλύτερος επενδυτής, οπότε θα πρέπει να τοποθετείται ο κλάδος για τις κινητές αξίες. Οπότε κάτι θα χάσουμε αν ακολουθήσουμε μια αυστηρά κλαδική τομεακή προσέγγιση. Επίσης ε, θα μπορούσατε να σχολιάσετε την ενίσχυση του συντονισμού που έχει προβλεφθεί ανάμεσα στου, στις, στους τρεις αυτούς τομεακούς οργανισμούς. Ο συντονισμός αυτός ε, είναι δυνατός από την ε, ισχύ του ίδιου του οργανισμού που συντονίζει και ακριβώς τι πώς συνδέονται αυτοί οι οργανισμοί με το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ηχέγγυα. Ε, ήμουνα στην Ουάσιγκτον ε, την περασμένη εβδομάδα με τον Πίτερ Σκίνερ και καλούσαμε θερμά τη ΕΙΠΑ να ε, εξάγουν τις εποπτικές τους δραστηριότητες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τόσο ώστε να υπάρχει ε, ισοδυναμία με τη φερεγγιότητα 2. Και τονίσαμε ότι Άμα υπάρχει μια ευρωπαϊκή ασφαλιστική εταιρεία και έχει μια θηγατρική και θεωρεί, θεωρηθεί από την Ομοσπονδιακή Αρχή ότι υπάρχει συστημικό κίνδυνο, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα και εμεί να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μα. Αυτό το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θέλουμε να είναι σε επαφή με το Συμβούλιο Σταθερότητα, όπω λέγεται, το αντίστοιχο όργανο στη ΣΥΠΑ. Αλλά α μην πέσουμε όμω την ίδια παγίδα, δηλαδή να παραγωνίσουμε την ασφάλεια. Μπορείτε να σχολιάσετε στο θέμα τη ενίσχυση αρχής του συντονισμού. Και κάτι άλλο ε, σχετικά με το ε, ε, επιτόκιο άνευ αν χρησιμοποιηθούν κρατικά ανάλογα α, μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλη πίεση γιατί ίσως μιλάμε αποκλειστικά για τη Γαλλία και τη Γερμανία και μπορεί να οδηγηθούμε σε στρέβλωση ή σε προκυκλικά φαινόμενα θα εσκύψετε σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, ε, γιατί ξέρω ότι ήδη ε, σας ε, το έχουν επισημάνει. Ευχαριστούμε για το πρώτο ζήτημα που θίξατε. Θεωρώ ότι υποδείξατε τη σωστή λύση, ενίσχυση του συντονισμού ανάμεσα στις συναρμόδιες αρχές, τους συναρμόδιους αυτούς οργανισμούς. Σήμερα αυτά που προβλέπονται στο τρίτο επίπεδο ε, ε, είναι ήδη θεμητά. Οι τρεις ε, οργανισμοί συνεργάζονται ήδη, συντονίζεται ο ρόλος τους με εγκάρσιο τρόπο και για τους τρεις τομείς δηλαδή και νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να είναι και το εφαλτήριο για την οικοδόμηση της νέας αρχιτεκτονικής. Εάν χρειαστεί άλλος οργανισμός που θα εποπτεύει τους άλλους τρεις, δεν νομίζω να προκύψει αυτό. Ε, δεν νομίζω να χρειαστεί η ενίσχυση του συντονισμού και ο σαφής προσδιορισμός των ρόλων τους ε, στην κείμενη νομοθεσία νομίζω ότι είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Για τις τεχνικές ε, διατάξεις και την έκπτωση, μιλώντας για το παθητικό, ο observe και το έχετε αυτό μέσα στο έγγραφο διαβουλεύσεων, έχει ορίσει μια σειρά κριτηρίων ε, για να δούμε αν ε, μια ε, βαθμολόγηση, ένας βαθμός είναι άνευ κινδύνου ή όχι. Μιλήσατε για τα κρατικά ομόλογα 3α. Αν δεν υπάρχει κανένας πιστοτικός κίνδυνος, πάρετε τα swap παραδείγματος χάρη ε, που ενέχουν ε, ε, κίνδυνο. τι θα κάνουμε, θα εξετάσουμε με βάση, την κατάσταση με βάση αυτά τα κριτήρια, αν συμφωνηθούν, και θα κάνουμε Προσαρμογέ για αυτά τα free rates, ε, τα επιτόκια άνευ κινδύνου, για να κατοχυρώσουμε ότι όντω είναι άνευ ε, κινδύνου. Ε, και θα συζητήσουμε με του εμπλεκόμενου φορείς για να βρούμε την σωστή λύση και το σημαντικότερο από όλα είναι να επιτύχουμε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ανταλλαγή απόψεών μας. Να είστε βέβαιος ότι θα είναι η πρώτη από πολλές ή από σειρά ανταλλαγών απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εκτενέστατες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις σας. Εγώ ευχαριστώ. No, no, we, we, Ευχαριστώ. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα μέχρι την επόμενη ε, ενότητα. Παρακαλώ αν αποχωρείτε τις αιθούσεις, αποχωρήστε τις ήχους. Κοινό σύστημα τώρα τη θέμα της αξίας, δεν είναι το επόμενο θέμα. Α, λάθος ημερήσια διάταξη ακολουθώ. Άλλοι έχουμε τώρα διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Αν θέλετε να βγείτε, βγείτε. Αλλά μην κάνετε φασαρία. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να μας παρουσιάσει το σημείο της. Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τέλη της προηγούμενης θητείας ενέκρινε μια σειρά νομοθετικών προτάσεων στα πλαίσια της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Μια κοινή στρατηγική και πρόταση οδηγίας για τη συνεργασία ακριβώς στη διοικητική στον τομέα της φορολογίας. Εγώ ως εισηγήτρια θα ήθελα να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και εδώ να τονίσω τη σημασία αυτού του νόμου και θα ήθελα να τονίσω τις βασικές πρόοδους ε, της ε, οδηγίας σε σχέση με τη σημερινή και την ισχύουσα δηλαδή. Μιλάμε ότι υπάρχει μεγάλη ε, φοροδιαφυγή που έχει ολέθριες συνέπειες ε, στους ε, κρατικούς προϋπολογισμούς και σε θέματα που είναι η παιδεία, η υγεία, η έρευνα, γιατί στερείται εσόδων το κράτος. Και επίσης παραβιάζεται και η αρχή της ε, φορολογικής ισότητας σε σχέση με τους μισθωτούς και τις εταιρείε. Και έχουμε και μεγάλη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Και αυτό επηρεάζει τη λειτουργία της αγοράς. Σε τέτοιους περιόδους λοιπόν με οικονομικής κρίσης όπου έχουν πολύ μεγάλα ελλείμματα τα κράτη-μέλη, η μείωση των εσόδων τους ε, ε, έχει επιπτώσει ακόμα πιο σοβαρές και πιο βαριές. Για να καταλάβουμε λοιπόν περί τίνος πρόκειται, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τον όγκο της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση κάποια στοιχεία είναι πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 200 δις και πλέον. Δηλαδή πάνω από, 20%, από 2% συγγνώμη, του ε, ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν δούμε τι γίνεται με την ανάκαμψη της οικονομίας και τι σχέδιο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί η οικονομική και η χρηματοπιστωτική κρίση, είναι το 1% σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, αν καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, αυτό ε, θα έχει μεγάλες επιπτώσεις και είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την ικανοποίησή μου στην, για την απάντηση του Επιτρόπου Κόβατς που θέλει να έχουμε περισσότερα μέσα και πιο αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη διοικητική συνεργασία. Ε, είναι διπλή η αιτιολόγηση αυτού, αυτής της ικανοποίησης. Γιατί ε, δεν διαταράσσεται η εσωτερική ε, φορολογική κυριαρχία των κρατών μελών, αλλά γίνεται συνεργασία διοικητική ε, με τρόπο πιο αποτελεσματικό για να μπορεί κάθε χώρα να διαχειρίζεται τα φορολογικά της. Επιπλέον, όσο προχωράει η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η οδηγία αυτή φαίνεται ότι είναι όλο και πιο απαραίτητη και πολιτικά και οικονομικά και διοικητικά και χρειάζεται σωστή φορολογική ε, προσέγγιση, αλλιώ δεν πρόκειται να λάβει σάρκα και ωστά το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η ισχύουσα οδηγία, επαναλαμβάνω, ήταν ένα καλό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τώρα ε, πρόκειται για ένα βήμα παραπάνω που δέχτηκαν σχεδόν όλα κρατημέλη. Και χρειάζεται νέα οδηγία, διότι η ισχύουσα δεν είναι πολύ συγκεκριμένη. Και υπάρχουν χώρες που θεωρητικά και επί της αρχής συμφωνούσαμε την οδηγία, τη στιγμή που έπρεπε να την εφαρμόσουν δεν έδειξαν τόσο μεγάλη προθυμία για να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι ότι έχει έρθει η στιγμή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να προχωρήσουμε σε νέα εργαλεία ε, φορολογικής συνεργασίας παράλληλα με την ολοκλήρωση της αγοράς. Υπό την έννοια αυτή η οδηγία που προτείνεται ε, σημειώνει ένα άλμα και ποιοτικό και ποσοτικό. Ποσοτικό διότι έχει νέα στοιχεία, νέες υποχρεώσεις και ε, ποιοτικό γιατί διευρύνει και βελτιώνει την ισχύουσα οδηγία. Χρειάζεται λοιπόν μια επιτάχυνση στην ε, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και είναι και επίκαιρο και λόγω της κρίσης διότι φάνηκε ακριβώς ποια είναι η εμβέλεια και το εύρος της ε, φοροδιαφυγής και πόσο αδιαφανής είναι η λειτουργία της αγοράς. Και όταν αυτά συμβαίνουν σε μία χώρα, βεβαίως καταλαβαίνετε ότι επηρεάζεται και αρνητικά και η οικονομία άλλων κρατών. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες και οι κυβερνώντες ότι υπάρχει ανάγκη πλέον να τερματιστούν σκανδαλώδεις καταστάσεις, όπως ε, ε, ζούμε τους τελευταίους καιρούς. Αν με επιτρέπετε θα σας έλεγα ότι τις μέρες αυτές και για λόγους δεοδολογικούς και ηθικούς και ε, οικονομικούς είναι απέτηση να μην χάνεται κανένα έσοδο, καμία πηγή εσόδων για την οικονομία μας. Γιατί ζούμε κρίση και χρειάζεται αντιμετώπιση της. δεν μπορεί το κράτος και οι εφορίες να μην έχουν τα έσοδα αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα για να ανακάμψει η οικονομία τους. Έρχομαι τώρα πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 1. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία που ισχύει σήμερα και μπαίνει και μια γενική ρήτρα που συμπεριλαμβάνει ε, για πρώτη φορά όλου του φόρου. Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας λοιπόν που θα αφορά όλους τους φόρους και τους άμεσους και τους έμεσους και τις υποχρεωτικές εισφορές στην ε, ε, κοινωνική ασφάλιση με εξαίρεση τους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ που είναι σε άλλη πιο προηγμένη οδηγία. Διευρύνεται λοιπόν το πεδίο εφαρμογή και είναι πρόοδο αυτό και είμαι πεπισμένη ότι η διεύρυνση θα αποτελέσει σημαντικό βήμα σε καλύτερη, μια καλύτερη φορολογική διαχείριση. Είναι σαφέ μήνυμα λοιπόν ότι ο ευρωπαϊκό μα ορίζοντα ε, στη διοικητική συνεργασία ε, σημαίνει κοινή ρύθμιση για όλου του φόρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγο για άμεση ανταλλαγή απόψεων ανταλλαγή συγγνώμη, προφοριών μεταξύ των διαφόρων φορολογικών αρχών. Οι εφορίε των κρατών μελών ε, θα επικοινωνούν μεταξύ του και θα ε, είναι και μέθοδο αναφορά αυτή. Εδώ είμαστε και πιο προηγμένοι ακόμα από τους ε, κανόνες του ΟΣΑ και από την οδηγία που ισχύει αυτόν τον καιρό και πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων στα τόπιν ετήσεως και μόνο και όχι αυτόματη στο ΕΚΟΦΗ αυτό το θέμα είναι ακόμα επίμαχο και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κατηγορηματικοί και να πούμε ότι υποστηρίζουμε αυτό το ποιοτικό άλμα, όπως σας είπα, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Βεβαίω. Θα πρέπει να βελτιώνεται όσο γίνεται ο τρόπος αυτός επικοινωνίας με την ανταλλαγή απόψε μεταξύ των φορολογικών αρχών ανάλογα με τις περιστάσεις και το είδος των στοιχείων που χρειάζεται και που ζητείτε κάθε φορά. Κεφάλαιο τρίτο ε, παρουσία στις διοικητικές έρευνες και συμμετοχή προσώπων υπαλλήλων φορολογικών αρχών από άλλα κράτη-μέλη. Με τη φυσική παρουσία δηλαδή υπαλλήλων. Συγκεκριμενοποιεί τη διαδικασία με λεπτομέρειες η νέα οδηγία και έτσι είναι πιο εύκολο να έχουμε ανταλλαγές υπαλλήλων η ε, αποστολή υπαλλήλων ε, μιας εφορίας σε ένα άλλο κράτος μέλος, βεβαίως όταν αυτό απαιτείται, ε, χωρίς να αφαιρεί τίποτα από τις εξουσίες και αρμοδιότητες των φορολογικών υπαλλήλων της λόγω χώρας. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι και η κατάργηση του τραπεζικού απορρίτου και καταραίει το βασικό εμπόδιο για τη διοικητική συνεργασία. Γι' αυτό στο κεφάλαιο 4 της πρότασης ρυθμίζονται οι όροι και οι υποθέσεις για να διαβιβάζονται οι πληροφορίες και τα έγγραφα ε, σχετικά. Είναι καινοτομία και είναι πάρα πολύ μεγάλο ε, επίτευγμα αυτό και θα έλεγα ότι είναι ε, ακριβώς και το, το αστέρι που ξεχωρίζει σε όλη την πρόταση οδηγίας. Μπορεί λίγες χώρες να, να διαφωνήσουν. γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία της οδηγίας αυτής, διότι σχεδόν ουσιαστικά υιοθετεί ε, τη σύμβαση του ΩΣΑ για τη φορολογία. Χρειάζεται καλύτερη φορολογική διακυβέρνηση και με συνεργασία ε, και σε αυτό έχει ε, δεσμευτεί και το G20 τερματίζοντας το τραπεζικό απόρριτο και αυτό είναι πάνδημη αίσθηση και αίτημα των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει και ένα μέτρο ε, μιας ρήτρας πλέον ε, ευνοημένου κράτους για να έχουμε προνομιακές σχέσεις με τρίτες χώρες και τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται ε, στα φορολογικά θέματα και με τρίτες χώρες. Τελειώνω. Τελειώνω λέγοντας ότι γενικά συμφωνώ με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι θεωρώ θετική. Βεβαίως χρειάζεται σε βάθος ανάλυση και θα κάνω και τροπολογίες για να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε ορισμένα στοιχεία της πρότασης αυτής. Είμαι στη διάθεσή σας ε, και των σκεδών εισηγητών για να συνεργαστούμε έτσι ώστε το κοινοβούλιο μας να εκφράσει την ανεπιφύλακτη και ε, ε, αναφυσβήτη υποστήριξη για να υπάρχει φοροδιαφυγή θα πρέπει αυτή να βρίσκει και πρόσφορο έδαφος για να ευδοκιμεί. Δηλαδή και θέλουν και μπορούν και θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε κάθε μέρα να είναι λιγότεροι εκείνοι που θέλουν και ακόμα λιγότεροι εκείνοι που να μπορούν. Σε δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να προχωρήσουμε, να περιορίσουμε τη δυνατότητα φοροδιαφυγής και να μην υπάρχουν και κίνητρα για τη φοροδιαφυγή. Να διατρανώσουμε λοιπόν προς τους πολίτες ότι είναι προτεραιότητα του Κοινοβουλίου κατά πολέμηση της φοροδιαφυγής και κάνει ό,τι μπορεί το Κοινοβούλιο για να την πετύχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εισαγωγή της Και ξέρετε και στη δική μου την έκθεση, στην προηγούμενη θητεία, με είχε υποστηρίξει για τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό. Οι σκιώδεις εισηγητές δεν μου έχουν, δεν είναι εδώ, δεν μου έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. κυρία Γκιούρι και αν έχουμε ακόμη λίγο χρόνο, θα πρότεινα να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Γκιόρη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την καλή διακυβέρνηση και προσπάθησα να μελετήσω αυτή την πρόταση και να τοποθετηθώ. Για την πρόταση Επιτροπής θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, για τα χρέη κτλ. Οπότε ε, το πρέπει να εφαρμόσουμε την ε, κείμενη νομοθεσία και να εμβαθύνουμε την συνεργασία των φορολογικών αρχών. Θα κάνω τρεις συγκεκριμένε ε, παρατηρήσεις για αυτήν την πρόταση. Πρώτον, πρέπει νομίζω να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στα είδη φόρων και τελών που προβλέπονται στην ε, ε, πρόταση της Επιτροπής για τα τέλη. Νομίζω ότι ο κανονισμός 515 του 97 τα καλύπτει. Δεν χρειάζεται άλλη νομοθεσία για τα τέλη αυτά. Μπορούν να αφαιρεθούν από αυτήν την πρόταση. Δεύτερη παρατήρηση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και για το ποιους τομείς πρέπει να καλύπτει αυτό το σύστημα αυτόματης ανταλλαγής. Νομίζω πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα διάφορα είδη εισοδημάτων και σε αυτή την οδηγία θα έπρεπε να προσδιορίσουμε και ένα όριο πάνω από το οποίο θα γίνεται αυτόματα η ανταλλαγή των πληροφοριών και αυτό σε κάθε τομέα. Τρίτον, προσπαθώντας να προσδιορίσουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι τομείς όπου θα ισχύει η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για τεχνικό ζήτημα δεν θα, ε, ήθελα να αποφασιστεί και να ρυθμιστεί με διαμέσου επιτροπολογίας. Ε, μέσα σε αυτή την οδηγία πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλα μέλη που έχουν ζητήσει το λόγο και στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μου πει μετά η εισηγήτρια αν θέλει να κάνει κάποια επιπλέον σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πρόταση αυτή εγγράφεται στα πλαίσια μιας σφαιρικής στρατηγικής την οποία καταθέσαμε το Μάιο του 2006. Ήσασταν εισηγήτρια εσείς τότε. Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει όλα τα μέσα διοικητικής συνεργασίας σε επίπεδο ΦΠΑ, σε επίπεδο άμεσης φορολογίας, το οποίο συζητάμε τώρα, και το θέμα της ανάκτησης ε, των χρεών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την πρόταση αυτή. Πάρα πολύ απλά η παρούσα οδηγία η οποία έγινε θα έλεγα το 77 δεν χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη εν και γι' αυτό θελήσαμε να την ενισχύσουμε. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενίσχυσης όπως το υπογράμμισε και η συγγήτριά σας. Πριν από τη διάλογο θα πρέπει να οργανωθεί η συνεργασία. Η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη δεν είναι οργανωμένη σε κοινοτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν όπως ακριβώς σε επίπεδο ε, δασμών και ε, ΦΠΑ προβλέπει να υπάρξουν κάποια γραφεία συντονισμού. Πρέπει επίσης να υπάρξουν εισαγωγές προθεσμιών για τις απαντήσεις στα αιτήματα, γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν ανταλλαγές πληροφοριών που καθυστερούν και δεν επιτρέπουν την καταπολέμηση της απάτης. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρξει πιο σύντομος χρόνος απάντησης. Η εισαγωγή επίσης εντύπων, διαδικασιών, τρόπων επικοινωνίας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν του ιδίου ε, τύπου θα έλεγα έγγραφα και η ενίσχυση του αυτόματου τρόπου ενημέρωσης. Γιατί επιμένουμε στον αυτόματο τρόπο ενημέρωσης, γιατί η ενημέρωση μετά από αίτημα που είναι το κατώτερο επίπεδο όσα αν θέλετε, ε, λειτουργεί άσχημα και λειτουργεί άσχημα γιατί υπάρχουν διαφορετικά στάδια. Ένα κράτος θα πρέπει να αποφασίσει να στείλει μια πληροφορία, να ζητήσει μια πληροφορία, ένα άλλο κράτος θα πρέπει να αποφασίσει να απαντήσει, και εν πάση περιπτώσει όταν έρχεται η ενημέρωση αργεί, καθυστερεί και πολλές φορές δεν έρχεται καν. Συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες καλύτερα, τα αυτόματα συστήματα ενημέρωσης και αυτό θα λειτουργήσει καλύτερα. Προβλέπεται επίσης και μια διαδικασία επιτροπολογίας η πρόταση αυτή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Συμβούλιο δεν θα έλεγα έγινε δεκτή από τα κράτη-μέλη, δεν θα υπάρξει επιτροπολογία παρότι εμείς είχαμε προτείνει κάτι τέτοιο. Εμείς θα διευρύνουμε λοιπόν τις προτάσεις αυτές για όλους τους φόρους εκτός από αυτούς όπου υπάρχει ένας κανονισμός. Η ρήτρα τώρα του ευνοούμενου κράτους. Είναι ένα καινοτόμο στοιχείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη αποδίδουν σε τρίτες χώρες καλύτερες μορφές συνεργασίας ενώ δεν το κάνουν στο ίδιο επίπεδο για τα κράτη-μέλη τα ίδια. Συνεπώς θελήσαμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τουλάχιστον ένα επίπεδο αντίστοιχο συνεργασίας και η κατάργηση του τραπεζικού απορρίτου θα έλεγα λόγω των τελευταίων εξελίξεων είναι κάτι το ίσον αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτη είχε προτείνει την κατάργηση του τραπεζικού απορρίτου εδώ και δεκαετίες. Σας ευχαριστώ. Θέλετε ξανά το λόγο. Κύριε Αλβάρες. Ευχαριστώ. Ε, είναι μακράς πνοή το θέμα αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Well, I'm, I'm sure. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα στο Κοινοβούλιο θα εκφράσουμε μια στεναρή γραμμή. Το χρονοδιάγραμμα νομίζω έχει ω εξή. 7 Δεκεμβρίου θα έχουμε την έκθεση. το έχει υποβάλει η ίδρυα. Και λίγο μετά θα λέγει η προθεσμία. 10 Δεκεμβρίου λέει εδώ προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, ενώ στι 7 θα φτάσει η έκθεση. Αυτό είναι το σημερινό χρονοδιάγραμμα, θα δούμε. Για να φτάσει στην Ολομέλεια μέχρι το Φεβρουάριο. Την πρώτη σύνοδο του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πάμε στο σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη που πολύ ε, πρόωρα υπερπίδησα. Τώρα είναι το κοινό σύστημα φόρου τη θέμενης αξίας και συγητής είναι ο Ούντο Μπούλμαν. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτό είναι διαβούλευση τώρα και ξανά μαζί της να κάνουμε μια έκθεση υπό το εξής υπόβαθρο άλλαξε σημαντικά το Συμβούλιο την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δική μας που είχαμε κάνει τότε αν θυμάστε στην έκθεση Ρωσάτη. Πρόκειται ε, για το δικαίωμα ε, παρακράτησης ε, προκατακτικής του φόρου και έχουμε μια επιφύλαξη σε σχέση με το Συμβούλιο και τη θέση του. Για κινητές αξίες, αν εφαρμοστεί τέτοιο μέτρο, μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλη αυθαιρεσία, διότι το Συμβούλιο αφήνει σε μεγάλο βαθμό τον ορισμό στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Και δεν μπορεί να υπάρχει ρύθμιση αξιόπιστη ε, για τους φορολογούμενους και για την οικονομία, για να υπάρχει και ένα στοιχείο συγκρισιμότητας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει ληφθεί υπόψη αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, η έκθεσή μας βασίζεται στην εξής ουσιαστική κεντρική ιδέα. Κάθε αλλαγή χρειάζεται μελέτη αντικτύπου και επιπτώσεων για να δούμε πού προκαλούνται ζημίες ή πού δημιουργείται κάποιο όφελος. Αυτό είναι το βασικό ε, σημείο της συζήτησης ε, ίσως και το επίμαχο, κατά τα άλλα συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μεγάλες ε, διαφωνίε σε σχέση με την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο το πρωί εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, τις εξαιρετικές σας υπηρεσίες. Πρώτης τάξεως είναι η γραμματεία. Ε, πραγματικά πρώτης τάξεως επεξεργασία του, του κ. Μπαρμπέρα και ευχαριστώ και όλους τους και για τη συνεισφορά τους. Μπορεί η έκθεση να είναι μικρή το θέμα μας, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Και σας ευχαριστώ για την καλή σας βούληση, για το πνεύμα συνεργασίας και την προσήλωσή σας για να μπορέσουμε τώρα να ε, έχουμε μια λογική πρόταση από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Φέρμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σύντομος θα σχετικά, παρόλο που το θέμα του φόρου τη θέμενη αξίας προσφέρεται να κάνει κανείς κάποια γενικά σχόλια. Αλλά αυτό το έχει εξεγγείλει για του χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια πρόγευση αυτή τη στιγμή να δούμε τι θα ζητηθεί για το ΦΠΑ. Υπάρχει πολλή δουλειά και ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με το ΦΠΑ και όχι σε τέτοιο επίπεδο μικρολογιστικής, ε, ένα στοιχείο, άλλο στοιχείο. Αν δούμε τι γίνεται ε, στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές, θα καταλάβετε τι Λυπάμαι που το Συμβούλιο δεν κατάφερε να συνεισφέρει θετικά να βοηθήσει να περιοριστεί λίγο αυτό το φαινόμενο. Έπρεπε να το πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένο με το Συμβούλιο. Ελπίζω του χρόνου να έχουμε μεγαλύτερη ευκαιρία αν τηρήσει τα επισημένα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω και το Συμβούλιο και προς το δικό του συμφέρον να παίξει και αυτό το ίδιο παιχνίδι. Γιατί εννοώ, τι εννοώ. Ε, προφανώς το Συμβούλιο ενδιαφέρει γιατί αυτά τα έσοδα πέρα από το μικρό βολό που πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στι έπες των κρατών μελών. Ο κύριος Μπούλμαν έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια με πολύ μεγάλη σκολασικότητα και ακρίβεια να κάνει την τροπολογία και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά την πολιτική μου ομάδα έδειξα καλή βούληση για να βάλουμε και εμεί το λιθαράκι μα να λυθούν τα προβλήματα και ελπίζω αύριο στην, ε, πλειοψηφία, στην ψηφοφορία συγγνώμη, να είναι μεγάλη πλειοψηφία και μια μικρή συνεισφορά από πλευρά μα. Προ το Συμβούλιο για να κινηθεί λίγο περισσότερο και να ακούει λίγο περισσότερο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τέτοια θέματα δύσκολα και κρίσιμα όπω είναι τα φορολογικά. Αχ, και αυτό έπρεπε να το πω. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη συνεργασία και ελπίζω να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα αύριο και προς το Συμβούλιο. Ένα κλάσμα, επαναλαμβάνω, είναι μόνο αυτό στο μεγάλο θέμα, στον ωκεανό ε, του ΦΠΑ που θα βρούμε μπροστά μας και θα συζητήσουμε το 2010. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όλοι Σμίτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Ούντο Μπούλμαν. Νομίζω ότι είναι λογική συμβαστική λύση που καταλήξαμε. Όπω είπε ο κύριο Φέρμπερ, ε, ε, μάλλον ε, αντίθετα με αυτό που είπε ο κύριο Φέρμπερ, δεν νομίζω ότι είναι σαφές το μήνυμα που περνάμε. Χρειάζεται κάποιε διευκρινίες στο κείμενο. Δεν ξέρω ποιο είναι ο σωστότερο τρόπος για να το κάνουμε, γιατί είναι τεχνικό το θέμα και υπάρχει η διάσταση ε, των απόψεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. στι τροπολογίε μου εγώ προτείνω το εξή. τουλάχιστον όταν τη συνέταξε τις τροπολογίες ε, αποσκοπούσαμε στο να διευκρινιστεί το κείμενο του Συμβουλίου. Καταλαβαίνω βέβαια και την, ε, το, τον κύριο Μπούλμαν ε, που επιχειρηματολογεί ότι χρειάζεται περισσότερη συζήτηση για να διευκρινιστούν αυτά τα σημεία που αναφέρω στις τροπολογίες μου. Υποστηρίζουμε την συμβαστική λύση και νομίζω ότι θα έχετε συντριπτική πλειοψηφία αύριο στην ψηφοφορία, κύριε Μπόλμαν. Ευχαριστούμε, κύριο Γκλουτ. Όχι, δεν έχετε ζητήσει το λόγο. Hans Peter Martin. Τα σοφά λόγια του ε, γείτονά μου ε, ε, προσβορά από τη Βαβαρία με κάλυψαν πλήρως και παρετούμε. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Um. Κάτι λέει ο κύριος Φέρμπερ, δεν ακούγεται. You Δεν έχει ζητήσει άλλο το λόγο. Κύριε Μπούλμαν, θέλετε να πείτε τίποτα, να ευθερολογήσετε και να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά, συνάδελφοι, έλεγα. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ρύθμιση συμφωνούμε και είναι πολύ ε, γρήγορη η διαδικασία. Κατά τα άλλα έχει δίκιο ο κύριος Φέρμπερ. Θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε ενεργητικά το θέμα. Στο μέλλον πώς μπορούμε να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα σε όλη την Ευρώπη για να μην έχουμε απάτες σε αυτά ε, τα εξωφρενικά ποσά και τα αστρονομικά που διαπιστώνουμε σήμερα στη διαφύγη. Ε, του ΦΠΑ. Και θα βοηθήσουμε όλοι και σίγουρα το Κοινοβούλιο δεν θα παρεμποδίσει τη διαδικασία. Δεν θα είναι το Κοινοβούλιο αυτό. Okay, thank you. I think that... Uh, Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ για αυτή η συζήτηση. Δεν ζητάει κανείς το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Λοιπόν, προχωρούμε. Αύριο θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Είναι το μόνο που έχουμε να πούμε. Το επόμενο θέμα είναι ε, το επαριθμό 6 της έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το έτος 2008. Εισηγητής είναι ο Έντουαρτ Σικλούνα. Um, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. which is in front of us um, in a very tight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 γιατί πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα οδηγήσει στην, σε μια αηφορία και στην οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Υπάρχουν διαφορές στην πολιτική που ακολούθησαν ορισμένες χώρες. Κάποιες χώρες επίσης σε επίπεδο χρεών και ελλημάτων είναι σε καλύτερη φάση από κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες έχουν και προβλήματα σε επίπεδο κόστους του εργατικού δυναμικού. Η Ευρωπαϊκή Ζώνη λειτουργεί ουσιαστικά σαν θα έλεγα η Ζώνη Ευρώ ενώ λειτουργεί σαν μια ομπρέλα περισσότερο και ε, όχι σαν κάτι ε, το διαφορετικό, σαν κάτι το αναγκαστικό και δεσμευτικό. Εμείς ε, συστήνουμε να ενισχυθεί ο διάλογος ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί αυτό βοηθά στον έλεγχο της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σχετικά με την ανεξαρτησία της ΕΚΤ, την οποία εμείς επιθυμούμε και θέλουμε να επιβεβαιώσουμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στις διαδικασίες διαβούλευσης για την επιλογή στελεχών και θα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία αυτή δίδοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγαλύτερο βάρος στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την επιβεβαίωση διορισμών που επιβεβαιούνται στην παρούσα φάση από το Συμβούλιο μόνο. Σχετικά με την Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου η οποία συζητήθηκε και σήμερα το απόγευμα. Οι κεντρικές τράπεζες και πολλοί παρατηρητές θεωρούν ότι δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ε, στα πλαίσια της διαδικασίας ορισμού του λεγόμενου συστημικού κινδύνου. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε τι εννοούμε με συστημικό κίνδυνο εφόσον θέλουμε να τον καταπολεμήσουμε. Και εφόσον θέλουμε να το καθιερώσουμε αυτό σαν ένα σημαντικό στόχο. Τέλος η έκθεση επιβεβαιεί και υπογραμμίζει το ότι η περιοχή του ευρώ έχει ενισχυθεί από την ύπαρξη του ευρώ και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει βοηθηθεί επίσης και από τις προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Uh, thank you. Mr. Ευχαριστώ κύριε Μπάλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον εισηγητή μας. Πολύ ισορροπή έκθεση και η πρότασή του. Δεν βλέπω να υπάρχει και ανάγκη για πολλές αλλαγές. Μερικά σχόλια και μόνο κάνω. Θα πρέπει να συζητήσουμε κιόλα. Ένα σχόλιο για το σημείο 2. Συγχαίρω για τη διορατικότητα του τον εισηγητή. Στο μεταξύ κυρώθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι θέμα που θα απασχολήσει την έκθεση του 2009. Για το σημείο 6 θα ε, έλεγα ότι να μην λέμε πολλές εμπορικές τράπεζες εδώ, many commercial ε, banks, αλλά να πούμε μερικές, a number. Το 7 είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητούμε έτσι εκτενέστατα. Εγώ νομίζω ότι η μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε γενικές γραμμές έχει γίνει σωστά. Κατά τα άλλα, ε, παγκοσμίω συνεννοείται η, τράπεζα με άλλες κεντρικές τράπεζες. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να την επικρίνουμε γι' αυτό. Να το συζητήσουμε παρακαλώ αυτό. Άλλη παρατήρηση. Στο σημείο 8, αντίστοιχα με το 6. Και εδώ δεν θα το γεννήκευα, δεν θα έλεγα οι τράπεζες, ορισμένες τράπεζες, όχι used by banks, used by some banks. Στο σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο συστημικός κίνδυνος δεν αυξήθηκε μόνο από την περιπλοκότητα της λειτουργίας. Είναι μία αιτία ε, από τις πολλές της κρίσης, γιατί αν υπήρχε διαφάνεια, αν υπήρχε καλή εποπτεία, που θα είχε αυξηθεί ε, όσο και η περιπλοκότητα των προϊόντων και των συναλλαγών, τότε θα ήταν πιο ε, ελέγξιμος ο κίνδυνος και θα είχε περιοριστεί. Για το 2013 νομίζω θα πρέπει η προσέγγιση μας να είναι λίγο πιο, διαφορετική. Ναι. Αυτό που ζητάτε είναι να συνεχιστούν τα προγράμματα ανάκαμψης ή μάλλον τα προγράμματα εθάρρυνσης και φορολογικών κινήτρων γιατί πολλά δεν έχουν αποδώσει αποτελέσματα αλλά προς το παρόν μέχρι να δούμε αποτελέσματα να μην προχωρήσουμε σε νέα προγράμματα. Αυτό άλλωστε πρεσβεύουν και οι Υπουργοί Οικονομικών. Στο σημείο 15 ε, θα πρότεινα να προσθεθεί μετά την τελευταία πρόταση ότι η αποτυχία να γίνουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις ε, θα ε, διακύβευε την αξιοπιστία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και γενικότερα το νόμισμά μας στο ευρώ καθώς επίσης και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχει να κάνει και θέματα με πολιτική απασχόληση και εργασία. Τελευταίο σημείο το 18 το είχα πει και στην ακρόαση τον κύριο Τρισέ, τον είχα ρωτήσει ήδη από την ακρόασή του. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να συμπεριληφθεί κάτι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζει και που δεν είναι να καταργεί την ανεξαρτησία της τράπεζας. Αυτό να το γράψουμε στο 18. Γενικά είναι καλή η πρόταση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή θερμότατα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια καλή δουλειά. Προετοιμάζουμε ορισμένες τροπολογίες για να βελτιώσουμε και να συμπληρώσουμε την έκθεση και θα ήθελα μέσα σε δύο λεπτά να μιλήσω για την εξωτερική διάσταση του Euro. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι σαν μέλη της Επιτροπής να ε, εμβαθύνει στο θέμα της εξωτερικής διάστασης του ευρώ γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το ευρώ είναι το πρώτο μεγάλο νόμισμα χωρίς κράτος πίσω του, ένα κράτος. Έχουμε φυσικά μια νομισματική ένωση και έχουμε ένα σημαντικό ομοσ... ομοσπονδιακό προϋπολογισμό αν θέλετε, αλλά το νόμισμά μας αυτό, το ευρώ παραμένει ορφανό δεν έχουμε επαρκή νομισματικό έλεγχο του ευρώ. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια προσωρινή αρχιτεκτονική ελέγχου, όπως είχε προβλεφθεί από τη συνθήκη του Μάστρεχ, τη συνθήκη της Λισαβόνας, διαφοροποιεί τα πράγματα. Η έξοδος από την οικονομική κρίση είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την οικονομία, αλλά προς το παρόν εμείς λόγω ακριβώς του υψηλού επίπεδου στο οποίο βρίσκεται σε, στις ισοτιμίες του ευρώ δημιουργεί προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα και στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν αναφορές στη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναφορές έλεγα στη νέα νομισματική αρχιτεκτονική γιατί το δολάριο θα εξασθενεί συνεχώς στο μέλλον, στο μέλλον και το γιουάν ε, ε, θα υποτιμάται μεν αλλά θα υποτιμάται με τεχνικό τρόπο, τεχνητό τρόπο και ε, στην ουσία θα έχουμε να κάνουμε με ένα νομισματικό dumping από πλευράς των Κινέζων, κάτι το οποίο ίσως μιμηθούν και οι Ρώσοι. Το ευρώ δεν ωφελείται και δεν εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες για να γίνει το ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο. Έχουμε ένα σαφές πρόβλημα μπροστά μας και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει επιτέλους κάποιες προτάσεις. Ευχαριστώ. Επίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή για το πρώτο σχέδιο της έκθεσής του Υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία χρειάζονται οπωσδήποτε ενημέρωση, λέει ο κύριος Γιανέπινγκ, ιδιαίτερα το σημείο 13, όπου ζητεί από τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τα μέτρα φορολογικών κινήτρων. Αν διαβάσετε τις εφημερίδες τις τελευταίες μέρες, βλέπετε ότι έχει εκτοξευθεί το χρέος 100% και πλέον του ΟΕΠ, ανάλογα με τη χώρα, και τα δημοσιονομικά ελλείμματα επίσης. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για να συνεχίσουμε πολύ περισσότερο με ε, τέτοια φορολογικά και δημοσιονομικά κίνητρα, γιατί ε, πραγματικά θα καλπάσουν προς τον όλεθρο τα δημοσιονομικά μας και οι προπολογισμοί. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ε, και πού είναι το μεγάλο κράτος πρόνοιας. Στο 14 δίνει λίγο μεγαλύτερη προσοχή στο χρέος ο εισηγητής λέει ότι αυτό από όσο είχαμε ε, προεξοφλήσει και όταν ξεπερνάει το 100% του ΑΕΠ το χρέος τότε και αν η ανάκαμψη οικονομία καθυστερήσει και έχουμε 1% περίπου αύξηση το χρόνο, δεν αρκεί αυτό για να αντιμετωπίσουμε το κόστος τη γύρανση σε πολλά κράτη-μέλη. Κινδυνεύουμε να έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Μετά γίνεται για το Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη. Θυμάμαι τη δεκαετία του 90 στην Ολλανδία μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που έλεγαν για τα κριτήρια ε, ότι ήταν ε, πραγματικά αποκρισταλωμένα, μετακίνητα, χαραγμένα σε μάρμα. Τώρα πού πάει το σύμφωνο σταθερότητας. Δεν ε, καλύπτεται, είμαστε σε έδαφος άγνωστο, δεν ξέρουμε προς τα πού πορευόμαστε και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από το υπηρεσιόδοξο τόνο και ύφος που αφήνεται στο ευρώ. Καλό το ευρώ και από την ομάδα μου, εγώ είμαι από εκείνους που είμαι υπέρ του, του ευρώ και έχω μεγαλώσει μέσα στο ευρώ. Αλλά δεν θα πρέπει να διακυβεύεται το ευρώ. Θα έχουμε στο μέλλον δυσκολίες και προβλήματα. Ένα τελευταίο αυτό που είπε και ο προηγούμενος ομιλητής η αξία και η δύναμη του ευρώ έχει πολύ μεγάλη σχέση ε, με τη μείωση της αξίας την υποτίμηση του δολαρίου. Ε, πριν από 15 μέρες είχαμε πάει στην Ουάσιγκτον και ευχαριστώ την πρόεδρο που μας προσκάλεσε να πάμε στη Federal Reserve και τους ρωτήσαμε τι γίνεται με την ανάκαμψη των ε, εξαγωγών. Κάνετε υποτίμηση του δολαρίου για να τονώσετε τι εξαγωγέ σα μαζικά και μα είπαν στη Fed ότι θα υποχωρήσει το, το ε, δολάριο σε επίπεδα αρχών του 2007 που ήταν 1,60 ευρώ. Εάν γίνει κάτι τέτοιο θα βρεθούν σε πολύ δινή θέση εξαγωγής Ευρώπης. Και εδώ σκέφτομαι τη Γερμανία που είναι ένα κράτος ε, το οποίο βασίζεται στην οικονομία του στις εξαγωγές και είναι και η κινητήρια δύναμη ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση. Χρειάζεται κάποια ενημέρωση σε σχέση με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Και καλό είναι να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, γιατί τα επόμενα 5-6 χρόνια το ευρώ θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μπερδέψει τα κουπιά. Άλλοι τρει ομιλητέ. Ε, Μποκρό, Μπόλμαν και Φερέρα. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Είναι πολύτιμη η έκθεση και για να μην μακρηγορήσω περνώ κατευθείαν σε κάποια λάθη που θα μπορούσαμε να διορθώσουμε παρόμο. Στο τμήμα, στο 7, υπονοείται με στην έκθεση ότι μπορεί η έκτη να έκανε λάθος που δεν μείωσε τα επιτόκια στο βαθμό που θα έπρεπε. Ταυτόχρονα στο 20 εκφράζει την ικανοποίηση διότι ε, έχει γίνει νόμισμα ε, σε ε, αποθεματικό νόμισμα σε διεθνές επίπεδο το ευρώ αλλά δεν γίνεται να τα έχουμε και τα δύο με στην ίδια έκθεση το ευρώ όπως είδαμε δεν υποστηρίζεται από ένα κυρίαρχο κράτος και από ένα κρατικό τομέα Οπότε πρέπει να είναι υψηλότερο το επιτόκιο ούτω ώστε να γίνει διεθνώς αποδεκτό αυτό το νόμισμα για ε, τα αποθεματικά. Και αυτή η κριτική στο 7 δεν αντιστοιχεί στα όσα συνέβησαν το 2008. Το μοναδικό λάθος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2008 ήταν που αύξησε τα επιτόκια τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Όχι ότι δεν ε, τα μείωσε επαρκώς. Δεν μιλάμε για το επίπεδο του επιτοκίου που έχει τη σημασία εδώ και μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ε, ως πρόβλημα. Άλλη ανακολουθία που θα ήθελα να υπογραμμίσω στην παράγραφο 6 εκφράζεται εδώ απογοήτευση διότι οι εμπορικές τράπεζες δεν έχουν μειώσει τα επιτόκια στο βαθμό που μείωσε το βασικό επιτόκιο η Μα Αυτό είναι φυσιολογικό γιατί επανατιμά το κίνδυνο όταν υπάρχει κρίση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θέλει οι εμπορικές τράπεζες ε, χωρίς να χρειάζεται να μειώνουν υπερβολικά τα επιτόκια γιατί σε περίοδο κρίσης ε, υπάρχει αυτό το λεγόμενο credit crunch ε, και δεν θέλετε να υπερτιμήσετε αυτά τα ενυπόθηκα δάνεια που έχουν δοθεί εκ των προτέρων από τις εμπορικές τράπεζες. Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα με την πίστη στη συνέχεια. Οπότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, καλά έκανε και άμβλυνε αυτόν τον κίνδυνο που ενέχουν τα υπερβολικά υψηλά επιτόκια των εμπορικών τραπεζών. Ξαναλέω, σε περίοδους κρίσης επαναξιολογείται ε, ο κίνδυνος από τις τράπεζες. Αυτό προβλέπετε. Ο κύριος Μπούλμαν. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Έτουαρτ Τσικλούνα για το πρώτο σχέδιο εκθεσής του για τη σαφή και ανάλυση και γλώσσα που χρησιμοποιεί για τις μακροοικονομικές εξελίξεις αλλά και για τις συστάσεις του και για το γεγονό ότι εκτιμά και τιμά την ε, νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η έκθεση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, στη συζήτηση του παλιού κοινοβουλίου, στο βαθμό που θυμάμαι και συμμετείχα εγώ, ε, στην Επιτροπή αυτή ήταν ένας χώρος όπου ακούγαμε διάφορες προτάσεις για το πώς θα πρέπει να κάνει κανείς νομισματική πολιτική και μάλιστα συγκρούονται αυτές οι απόψεις και ποτέ δεν κάναμε αυτό που θα ε, έπρεπε, αλλά προτιμούσαμε να αναφέρει ο καθένα την αγαπημένη του προσέγγιση. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είμαστε σε περιόδους κρίσης που δεν μας επιτρέπουν τώρα να κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις και ε, ο καθένα να βάζει τις απόψει του σε μια τέτοια έκθεση. Δεν ε, χωράνε τώρα τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να βρούμε κοινό έδαφος και να πούμε ε, σε αυτό το όργανο της Ένωσης τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς ε, είμαστε το μόνο σοβαρό όργανο ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας και δεν έχουμε μόνο το δικαίωμα, έχουμε και το καθήκον και την υποχρέωση να λέμε και να διατυπώνουμε τις προσδοκίες μας παρακαλώ και εύχομαι όλοι οι συνάδελφοι και όλοι οι και άλλοι που θέλουν να κάνουν τροπολογίες να μην αποδυναμώσουν την άποψη του εισηγητού. Αν θέλετε να βοηθήσετε να ενισχυθούν κάποια στοιχεία, να ενημερωθούν κάποια στοιχεία, να βελτιωθούν όπου αυτό απαιτείται. Αλλά παρακαλώ μην μπείτε στον πειρασμό να πέσουμε σε μια γενική ε, τοποθέτηση και να βγει ένα κείμενο σούπα που το κοινοβούλιο να μην έχει τίποτα να πει. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους τομείς όπου λόγω του θεσμικού μας ρόλου πρέπει να ε, απευθυνθούμε στην τράπεζα. Ε, στα σημεία 17 και 23 θα πρέπει να βοηθήσουμε να ε, βγουν σωστά προς τα έξω για να είναι σοβαρή φωνή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Είναι απέτηση των καιρών αυτή και η έκθεση πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ. Ελίζα Φερέιρα. Thank you very much. Well, Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον εισηγήτη για αυτό το σχέδιο έκθεσης που είναι πλήρως σοσκελισμένο. Θα συμφωνήσω με τον Ούντο Μπούλμαν. Αν είναι να ενισχύσουμε κάποιο τύχη, θα πρότεινα να διασαφίσουμε τη διατύπωση στο 23. Η διεθνής θέση του Euro, του ευρώ, στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας πρέπει να οροθετηθεί με ακρίβεια και να περάσουμε ένα σαφές μήνυμα σε αυτό το τομέα. Τι συμβαίνει. Ο ρόλος του ευρώ σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο και το νόμισμα της Κίνας δημιουργεί ανισορροπίες ως προς επιπτώσεις που έχει στην πραγματική οικονομία στην Ευρώπη αλλά και σε επιμέρους χώρους ανάλογα με με το αν η πραγματική οικονομία προσανατολίζεται προς τις εισαγωγές ή προς τις εξαγωγές. Θέλω να τονίσω αυτό το σημείο, διότι δείχνει την στενή σχέση που υπάρχει, που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην ΟΝΕ και στην πραγματική οικονομία ε, των χωρών της ζώνης ευρώ. Θα ήθελα να το λάβετε αυτό υπόψη όταν εξετάζετε τις τροπολογίες που υποβάλαμε. Αλλά μην, ξεχνάω μην ξεχάσω να σας αποδώσω τα εύσημα για αυτά που ήδη έχετε καταφέρει. Πρόεδρος, ε, είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση για το ευρώ και ένα αποθεματικό νόμισμα και τι πρέπει να κάνουμε. Θα θέλατε να κάνετε κάποια καταληκτικά σχόλια, κύριε Σίγητα. Πέντε λεπτά. Έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ για αυτά τα σχόλια. δύο εξαιρουμένων ε, με βρίσκουν σύμφωνο κυρίως αυτό που είπε ο κύριος Μπούλμαν ότι θα πρέπει να ε, διευκρινίσουμε τη διατύπωση σε κάποιες παραγράφους χωρίς όμως να αλλοιώσουμε το νόημα. Ε, ξέρετε, σε κάποιες προηγούμενες εκθέσεις έχουν γίνει, έχει γίνει ακατάληπτο το κείμενο λόγω των πολλών τροπολογιών. Αν το έχουμε αυτό κατά νου. Θα αρχίσω από το τέλος. Παράγραφος 23. Ε, Τονίζεται εδώ η ενίσχυση του ρόλου του ευρώ, όχι η ενίσχυση του ευρώ. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν θέλω να είναι ισχυρό το ευρώ ώστε να πλήξει την ανταγωνιστικότητά μα σε μια περίοδο που πρέπει να εξάγουμε περισσότερο. Αλλά αν ο ρόλος και η σταθερότητα που ε, ο ρόλος ενός νομίσματος ε, ε, διαφέρει από τη σταθερότητα ενός νομίσματος. Πρέπει να κάνουμε αυτή την διάκριση, ούτω ώστε να μην δημιουργηθεί σύγχυση. Κύριε Μπάλτσε, το είπατε καλύτερα και από μένα. Φυσικά μπορούμε να επιφέρουμε όλες αυτές τις χρήσιμες αλλαγές στο κείμενο. Για τα φορολογικά κίνητρα και πολλοί συναδελφοί σχολίασαν αυτό το ζήτημα Άλλο να αυξήσουμε τα φορολογικά κίνητρα και άλλο να τα διατηρήσουμε. Και η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας παροτρύνουν να συνεχίσουμε όταν βλέπουμε σημάδια ε, ε, βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και προσεκτικοί διότι δεν θέλουμε οι χώρες, οι φορολογούμενοι, μελλοντικές γενναίες να επιβαρυνθούν με δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσια χρέη που το μόνο που θα κάνουν είναι να ε, πλήξουν τις ε, οικονομίες που ακολουθούν αναπτυξιακή πορεία. Θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τους συναδέλφους και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω εγώ τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. Ξέχασα την κυρία Γιώρη. θέλετε να κάνετε ερώτηση. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη που σας ε, ξέχασα. Ε, μπορούμε όμως να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα στη μέσα διαταξή που είναι έκθεση για το 2009, ετήσια δήλωση για την Ευρωζώνη και τα δημόσια οικονομικά πρώτη ανταλλαγή απόψε. Η συζητής είναι ο Σβέν Γκίγολτ. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Ακόμα και αν υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί αγενές να μιλάει κανείς γερμανικά. Είχαμε μια μικρή ανταλλαγή εύθυμη προηγουμένως. Επιτρέψα μου λύσω τη γλώσσα μου γιατί μπορώ να εκφραστώ με μεγαλύτερη ακρίβεια. Λοιπόν, και αυτή η έκθεση έχει σημασία για την ετήσια δήλωση δηλαδή για τη ζώνη του ευρώ και τα δημόσια οικονομικά. Εδώ παρουσιάζονται κάποια στοιχεία που δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά και χαρμόσυνα. Δηλαδή, παραμένουν πολύ δυσμενείς οι εξελίξεις και οι διαδικασίες. Αν δείτε και τις φθινοπορεινές προγνώσεις, παραμένουν χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που προβλέπονται και για το επόμενο έτος και χαμηλή ανάπτυξη και χαμηλό δυναμικό με τα αντίστοιχα αποτελέσματα και επιπτώσεις και για τα δημόσια-οικονομικά και για την απασχόληση. Επιπλέον, θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ύπαρξη του ευρώ, όπως και η νομισματική πολιτική και η επεκτατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και η επεκτατική φορολογική πολιτική οδήγησε στο να μην μας πλήξει ακόμα βαθύτερα η κρίση. Αυτό έχει σημασία και θα πρέπει να το σκεφτούμε στην ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε στη συνέχεια. Και η κρίση κατέδειξε και ορισμένες αδυναμίες της οικονομικής διακυβέρνησης και της δομής της Ευρωζώνης και της νομισματικής αλλά και της οικονομικής ένωσης. Αυτό φαίνεται και στις εκθέσεις ε, που μας παρουσιάζουν για τα δημόσια οικονομικά και με τρόπο σαφή. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε αυτό. Βλέπουμε ανισορροπίες εσωτερικές και εξωτερικές. Οι εσωτερικές ποιες είναι. Είναι ότι ορισμένες ε, εξελίξεις ε, μισολογικές ας πούμε και τα ισοζύγια τραχουσών συναλλαγών και τα εμπορικά ισοζύγια διαφέρουν. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές και, μέσα και προς τα έξω. Έχουμε μεγάλες ανισορροπίες μεταξύ των διαφόρων ε, νομισματικών ε, ζωνών, αλλά και το 2008 είδαμε πολύ μεγάλους κραδασμούς με υψηλές τιμές ε, των πρώτων υλών και της ενέργειας. Κάτι άλλο που αναφέρει επίσης μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι ε, αδυναμίες στη ρύθμιση και στην εποπτεία των χρηματαγωγών. Θεωρώ βέβαια ότι αυτό το ζήτημα δεν θα μας απασχολήσει στην παρούσα έκθεση. Υπάρχουν άλλες διαδικασίες και άλλα κείμενα που το διαπραγματεύονται σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να πω κι εγώ σε αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αδυναμίες στον συντονισμό της φορολογικής πολιτικής και στο παρελθόν αυτό ε, έδειξε μεγάλες τάσεις κυκλικών ε, φαινομένων, παράλληλα με τους κύκλους δηλαδή της οικονομίας και θα πρέπει να δούμε πώς για να βγούμε αυτή την κρίση πώς θα συντονιστούμε φυρολογικά. Εγώ θα πρότεινα να αναφερθούμε λιγότερο στην έκθεσή μας και στην νομισματική πολιτική γιατί έχουμε την προηγούμενη έκθεση οπότε θα κερδίσουμε και χώρο για να αφιερωθούμε αλλού. Ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα για το ρόλο του ευρώ ε, και τα εξωτερικά προβλήματα που συνδέονται με αυτό. Δηλαδή η ισοτιμία του ευρώ με τα άλλα μεγάλα διεθνή νομίσματα. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο στην έκθεση όμως που αναφέρεται στο ευρώ. Τώρα, αν θέλετε να περάσουμε στις λύσεις για τα προβλήματα τα οποία έχουμε αναγνωρίσει και εντοπίσει γιατί η κρίση τα κατέστησε ιδιαίτερα ορατά, Υπάρχουν ορισμένα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στη διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης και να τα συζητήσουμε σε βάθος. Να μην τα επαναλάβω εγώ, αλλά υπάρχει έκθεση Μπερές που είναι εκτενής ε, για ε, τα 10 χρόνια ζωής του ευρώ. Και εκεί η κυρία Μπερές έκανε μια σειρά συστάσεων. Σε αυτές θα πρέπει να επανέλθουμε στο βαθμό που δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα ή δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, απλώς να θέσω υπόψη σας ορισμένα ζητήματα που έχουν σημασία μακροοικονομικά. Ένα. Τι μελγενέστε με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο χρέωσης όπου οι κανόνες του συμφώνου δεν έλαβαν αρκετά υπόψη αυτό το γεγονός. Προφανώς γιατί τότε δεν ε, ε, θεωρεί το αυτό από κανένα ούτε επιθυμητό ούτε πιθανό ότι πρόκειται ποτέ να προκύψει. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Οι κανόνες που έχουμε για την εξόφληση του χρέους ε, δεν επαρκούν και θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα επανέλθουμε σε επίπεδα βιώσιμα. Το ίδιο ισχύει ε, ε, για τις μεγάλες εσωτερικές ανισορροπίες που σας έλεγα προηγουμένως και πώς θα αντιμετωπίζονται αυτές. Θα πρέπει να το συζητήσουμε εδώ σοβαρά αυτό. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μήπως θα πρέπει να ε, βάλει και μια εξωτερική διάσταση πέρα από το δημόσιο χρέος και τα δημόσια ελλείμματα που να δίνει κίνητρα σε κάποιες χώρες που έχουν μεγάλα πλεονάσματα να μειώσουν τα πλεονάσματά τους και να δίνει και μεγάλα κίνητρα σε χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα να μειώσουν και αυτές τα ελλείμματα τους. Άλλο θέμα. Πώς συντονίζουμε περισσότερο τη φορολογική μας πολιτική και πώς θα καταφέρουμε οι συμφωνίες που υπάρχουν καταρχή ε, να έχουν και αυτά αποτελέσματα, να εφαρμόζονται στην πράξη δηλαδή και εδώ χρειάζονται απαντήσεις. Εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο εξή. Αν δούμε την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και τη συγκρίνουμε μεταξύ τους, τι ε, έδειξε η κρίση ότι διαφέρουν τα επιτόκια στον δανεισμό για την αντιμετώπιση του χρέους. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε πλέον ότι ε, οι χώρες μόνες τους θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτό το πρόβλημα. Ακόμα και αν είναι το κύριο καθήκον τους, το κάθε κράτος θα πρέπει να τηρεί τα δημόσια οικονομικα του σε υγιή επίπεδα. Ωστόσο, θα πρέπει να προβληματιστούμε, να δούμε πώς χρειάζονται ευρωπαϊκοί μηχανισμοί και ποιοι θα είναι αυτοί για να βοηθήσουμε τα μεμονωμένα κράτη-μέλη να εξηγιάνουν τα δημόσια-οικονομικά τους. Επανέρχομαι στην έκθεση Μπερές Λάγκεν που προτείνει ευρωομόλογα. Αν γίνει σωστά αυτή η προσπάθεια Ποιο είναι το σκεπτικό. Οι χώρε εκείνες που πρέπει να, ψηλών, να πληρώνουν ψηλά επιτόκια ε, για να δανείζονται για να καλύψουν το έλλειμμα, θα πρέπει αυτό το ποσοστό σε αλληλεγγύη ε, να ε, ε, το μοιράζονται με χώρες που έχουν χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού. Αυτά είναι κίνητρα για την εξηγίαση του προπολογισμού των κρατών και των δημοσίων οικονομικών. Επαναλαμβάνω, ε, το ευρωπαϊκό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα φορολογικής διακυβέρνησης δεν βοηθάει πάρα πολύ για να συλλέγονται οι φόροι στην πραγματικότητα. Προηγουμένως συζητήσαμε για την απάτη στο ΦΠΑ, η συνεργασία για τους άμεσους φόρους, ιδιαίτερα ε, τους φόρους από ε, έσοδα κεφαλαίου με τις διάφορες μορφές. Οπότε και εδώ τίθεται το θέμα ε, της κοινή φορολογικής βάσης και ε, φορολογικοί συνεργαστές αλλά και οι νέες πηγές εσόδων όπως η φορολόγηση της ρήπανσης του περιβάλλοντος ή η φορολόγηση των ε, χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών. Τέλος, στην έκθεσή μας θα πρέπει να λάβουμε θέση για μια συντονισμένη στρατηγική εξόδου από την κρίση και από την ε, επεκτατική φορολογική ε, πολιτική. Και εκεί συμφωνούν οι περισσότεροι οικονομολόγοι ότι η νομισματική πολιτική μπορεί να παραμείνει έτσι, επεκτατική σε μεγάλο χρονικό διάστημα ε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην γίνουν αυτά βεβαιασμένα και πολύ νωρίς, ε, όπως άλλωστε συζητάει και το ΕΚΟΦΗΝ. Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι πώς θα περάσουμε γρήγορα σε εξυγίανση του προπολογισμού, αλλά πού θα βρούμε πηγές για νέα ε, δυναμική που να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, που να δημιουργούν και επενδύσεις γνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι ο πλανήτης είναι περιορισμένος και η κλιματική αλλαγή σοβαρή και χρειάζεται και σοβαρή αντιμετώπιση. Και τώρα το τελευταίο, θα ήθελα να κάνουμε εδώ μια ειλικρινή συζήτηση, να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πολλά κράτη-μέλη, ιδιαίτερα τα κράτη της Βαλτικής, αλλά και άλλα, και η Πολωνία, είπαν ότι θέλουν να μπουν στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν αυτό τον καιρό κυρίως στη Βαλτική, πώς ε, αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα ε, της επιθυμίας ένταξης στην Ευρωζώνη, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα σημαίνει και μεγάλες ενισχύσεις για περισσότερη σταθερότητα στις χώρες αυτές. Θα πρέπει τα κριτήρια να είναι άκαμπτα, σκληρά, που έτσι κι αλλιώς δεν τα πληρούμε εμείς στο εσωτερικό της Ευρωζώνης είναι σκόπιμο να διατηρηθούν αυτά. Και αυτό το θέτω προσυζήτηση. Έκανα πολλέ ερωτήσει. Περιμένω να δω τι θα πείτε κι εσείς, να ακούσω τις απόψει σα και ευχαριστώ για τις συζητήσεις που είχαμε ήδη με τους σκιώδες ηγητέ. Τουλάχιστον για μένα ήταν πολύ διαφωτιστικές. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Chers collègues, bonjour. Euh, je tiens... Καλημέρα συνάδελφοι να ευχαριστήσω τον κύριο Γκίγκολτ. Είμαι εισηγήτρια για την ομάδα μου, σκιώδης εισηγήτρια δηλαδή για το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας κύριε εισηγητά. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι αρκετά αντικειμενική. Κάποιες παρατηρήσεις όμως, επί των οποίων νομίζω ίσως να υπάρξει μια συζήτηση για την ανεργία. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται πάρα πολύ συνοπτικά στην ανεργία. Ενώ είναι ένα από τα βασικά θέματα, να μην πω το πιο βασικό θέμα που έχουμε μπροστά μας και πρέπει να λύσουμε στην Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το επίπεδο. Φτάνει το 10% στη ζώνη ευρώ κατά μέσον όρο και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να εγνοήσουμε για, για τα χρέη των κρατών. Επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάγνωση την οποία κάνει, δηλαδή ότι υπάρχουν, υπάρχουν υποχρεωμένες χώρες, αλλά δεν κάνει και πάρα πολλές προτάσεις και δεν προτείνει ιδιαίτερες λύσεις για τη μείωση αυτής της υπερχρέωσης. Νομίζω ότι είναι ένα τομέα στον οποίο πρέπει από κοινού να εργαστούμε για να δούμε τι μέσα μπορούμε να φανταστούμε για να χρησιμοποιήσουμε για την καταπολέμηση της υπερφρέωσης και τι μέσα μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας για να υπάρξει μια ουσιαστική, μια δυναμική οικονομική ανάκαμψη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εντάξουμε στην έκθεση. Πρέπει επίσης στα πλαίσια της έκθεσης αυτής να ξεκινήσει μια σαφέστατη συζήτηση σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την θα έλεγα δυνατότητα που έχει σήμερα να νομιμοποιείται και να επηρεάζει την Ευρωζώνη. θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάποιες δυνατότητες συνεργασίας, αν και δεν προβλέπονται θεσμικά, και για τα ευρωομόλογα, για την οικονομική συνεργασία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο του Eurogroup. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την θέση της Ευρώπης αυτόνομα στο εσωτερικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν και να απαντηθούν. Ευχαριστώ. Κύριε Θα πρέπει να σταθούμε λίγο στη διάγνωση την οποία κάνει η έκθεση αυτή, ότι δηλαδή η κρίση αυτή δεν είναι μια απλή χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία να οφείλεται αποκλειστικά στην, θα έλεγα, ελαφρώμια λιστάση των τραπεζών που επηρέασε την πραγματική οικονομία. Η κρίση ρευστότητας σημειώνεται για πρώτη φορά στη ζώνη ευρώ τον Οκτώβριο του 2008 ενώ οι μακροοικονομικές ανισότητες της ζώνης αυτής εμφανίζονται πολύ νωρίτερα και ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2008 αντιστρέφεται η συγκυρία και οι περισσότερες από τις χώρες της ζώνης ευρώ περνούν σε αρνητική ανάπτυξη πριν από την κρίση ρευστότητα του Οκτωβρίου το δεύτερο τρίμηνο του 2008. Και για τη ζώνη ευρώ πιο συγκεκριμένα, στις δύο κινητήριες δυνάμεις αυτής της ζώνης, Έχουμε μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε πλεονασματική αποτεμίευση με μια χρηματοπιστωτική αγορά η οποία υποφέρει διότι μειούται η επένδυση και η κατανάλωση σταματά πλέον και δεν είναι ο βασικός κινητήρας ανάπτυξης. Η ίδια η Γερμανία που ήταν καλή στις εξαγωγές θα υποστεί τις συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης και γνωρίζετε ότι φέτες θα έχει μια αρνητική ανάπτυξη που θα φτάνει το μείον 5. Υπάρχουν λοιπόν παράγοντες που θα πρέπει να εντοπιστούν, παράγοντες μακροοικονομικής ανισότητας. Εφόσον πράγματι θέλουμε εμείς να διαμορφώσουμε τις σωστές πολιτικές εξόδου από την κρίση. Εγώ άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τον κύριο Αλμούνια την προηγούμενη εβδομάδα και εξεπλάγην. Εξεπλάγην διότι ομιλούμε για μια πολιτική εξόδου από την κρίση υποθέτοντας ότι θα πρέπει να αυστηροποιήσουμε τη δημοσιονομική πολιτική και ίσως και τη νομισματική πολιτική από το 2010. 2011 μάλλον. Αυτό σημαίνει ότι από τον επόμενο Οκτώβριο του 2010 οι συνάδελφοί μας θα ασχοληθούν με προϋπολογισμούς οι οποίοι θα θεωρούνται ε, θα έλεγα κυρίαρχα λυτοί τι μας λέγουν όμως οι προβλέψεις των μακροοικονομολόγων. Ότι η μακροοικονομική κατάσταση του 2010 στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγήσει σε έναν αριθμό ανάπτυξης που θα κινείται περίπου στο 0,5%. Όπως το είπε η προηγούμενη συνάδελφος, έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό στην ανεργία. Ξέρουμε ότι κάτω από 1,5% ρυθμό ανάπτυξης θα καταστρέφονται συνεχώς θέσεις απασχόλησης. Αυτό οφείλεται στο ότι η δυνατότητα χρήσης του παραγωγικού δυναμικού είναι πάρα πολύ χαμηλά στη Γαλλία και τη Γερμανία, κάτω του 70%. Και με τέτοιου είδους χαμηλά επίπεδα, στην ουσία βρισκόμαστε σε μια υποβαθμισμένη χρήση των παραγωγικών δυνατοτήτων, ως εκ τούτου η λιτότητα δεν θα βοηθήσει. Θα ήταν λοιπόν λάθος να πιστέψει κανείς ότι ήδη από το 2010 θα πρέπει να εμπλακούμε σε πολιτικές οι οποίες είναι συμβατές με μια κατάσταση πλήρους απασχόλησης αλλά πλήρως ακατάλληλες με μια κατάσταση ανεργίας. Πρέπει λοιπόν να το πούμε αυτό και να το υπογραμμίσουμε στην έκθεση. Αυτό να ξεκινήσει συζητήσεις και σε άλλες εκθέσεις. Μιλήσαμε πολύ για τα χρέη. Εγώ θα είμαι υπεύθυνο ε, για ε, τα δημοσιονομικά και τελειώνω εδώ για να μην μακρηγορώ, όταν λέμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί μια κάποια δυναμική ανάκαμψη ήδη από τον επόμενο χρόνο. Κάτι δηλαδή το οποίο να ξεπερνά το σύμφωνο σταθερότητας γιατί βρισκόμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση ύφεση, το οποίο περιγράφεται θα έλεγα σαν φαινόμενο ε, το 2005 σε μια κατάσταση όπου η ανάπτυξη είναι κάτω του ρυθμού του 2%. Κάτω από τις συνθήκες αυτές είναι δυνατόν επίσημα και νόμιμα να κρατήσουμε ελλείμματα δημοσιονομικά μεγάλα για να υποστηρίξουμε την οικονομία. Δεν είναι εκεί όμως η συζήτηση υπάρχουν ε, θα έλεγα καλά ελλείμματα και κακά ελλείμματα και θα πρέπει να τα εντοπίσουμε αυτά τα καλά και κακά ελλείμματα. Καλά ελλείμματα είναι όταν υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη, όταν δηλαδή πετυχαίνονται οι στόχοι των προϋπολογισμών και υπάρχουν και κακά ελλείμματα όταν οι στόχοι τους οποίους καθορίζουν και αναζητούν να πετύχουν οι προϋπολογισμοί δεν επιτυγχάνονται. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν στις διάφορες χώρες τα καλά και τα κακά τέτοιου είδους ελλείμματα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι έχουν ζητήσει άλλα μέλη το λόγο. Σας ευχαριστώ. Είχαμε μια ανοιχτή συνάντηση των συντονιστών με τον Επίτροπο Αλμούνια, αλλά επειδή καθυστέρησε η δημοσίευση της έκθεσης αυτής, μετά και από την τελευταία παρέμβαση καλό θα είναι να μας πει και ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής της Αρμόδιας το που βρισκόμαστε σήμερα. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας και αν πάρετε λίγα λεπτά από τον χρόνο αυτό θα επανέλθω στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Μια ερώτηση. Ε, θέλετε να σχολιάσω και την έκθεση για τα δημοσιοοικονομικά ή μόνο για την ετήσια έκθεση για το 2009. Είναι συνδυασμένα τα δύο ζητήματα στη δική μας την έκθεση, οπότε ό,τι θέλετε. Αλλά μη μακρηγορήσετε υπερβολικά. Όχι, όχι, θα είμαι σύντομος. Έχετε όλη την έκθεση εξάλλου. Ε, σας την έχουμε στείλει. για την ετήσια έκθεση για τη ζώνη ευρώ είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ως follow-up της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην οποία αναφέρθηκε ο εισηγητής. Για μας η ετήσια έκθεση είναι σημαντικό στοιχείο για να ενισχύσουμε το διάλογο με το Κοινοβούλιο για όλα τα ζητήματα που άπτονται τη ζώνης ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό δεδομένης της κρίσης ε, και του follow-up αυτής. Ε, τα βασικά μηνύματα φαίνονται στην ετήσια έκθεση ε, η κρίση έχει αφήσει κάποια δυσεπίλητα ζητήματα μετά από την πρώτη επιτυχή δεκαετία της ΟΝΕ η κρίση επίσης ε, έδειξε όλες τις ανισορροπίες που υπάρχουν στη ζώνη ευρώ και είδαμε ότι είναι πιο ευάλωτα κάποια κράτη-μέλη σε σχέση με άλλα. Τα εκκρεμή ζητήματα σχετίζονται επίσης με την δυνατότητα αντίδρασης της ζώνη ευρώ ε, για ε, μια τέτοια κρίση και είδαμε ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματική η ζώνη ευρώ όσο περιμέναμε. Ακούσαμε διάφορα άλλα στοιχεία, τον κατακαιρματισμό της εποπτείας, ε, η έλλειψη ε, δυνατότητας διαχείρισης της κρίσης σε κάποιες χώρες της ζώνης ευρώ, επίσης ε, κατάσταση των δημοσιοοικονομικών στο παρελθόν και γενικότερη δομή διακυβέρνησης που πρέπει να αναβαθμιστεί. Τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Ε, η δήλωση τονίζει, ε, πανέρχεται μάλλον, σε μηνύματα κλειδιά ε, που υπήρχαν στην περσινή έκθεση ένα βασικό στοιχείο είναι η αποτελεσματικότητα της ε, χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Ε, χρειάζεται διεύρυνση και εμβάθυνση. Διεύρυνση διότι πέρα από τις εξελίξεις, ονομαστικούς δείκτες, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις ως προς την ανταγωνιστικότητα και τις εσωτερικές εξελίξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε ε, κάποιες συγκεκριμένες των χρηματοπιστωτικών αγορών για να χειριστούμε την ε, κρίση. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πρόκληση ως προς τον συντονισμό για αυτή την στρατηγική εξόδου για τα δημοσιοοικονομικά στη ζώνη ευρώ. Χρειάζεται πιο εντατικό συντονισμός, αυτό φαίνεται έκδηλα μέσα στην έκθεση, και έχουμε επίσης την εντύπωση ότι υπάρχει περιθώριο ελιγμών για την ομάδα ευρώ ε, για να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο που πρέπει να έχει στη ζώνη ευρώ. Ακούγοντας ε, τις ερωτήσεις ε, ε, για την δομή της έκθεσης βλέπουμε ότι γίνονται κατανοητά τα βασικά ζητήματα. Μία έκκληση από πλευράς μας τώρα σε σχέση με την δυναμικότητα, την αυξανόμενη δυναμικότητα της G20 ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να σκέψει στο θέμα της εξωτερικής εκπροσώπησης ε, και να αποδώσει τη δέουσα σημασία σε αυτό το ζήτημα. Για την έκθεση για τα δημοσιοοικονομικά θα ήθελα να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Η φετινή έκθεση δείχνει πώς αντιμετώπισαν την κρίση τα κράτη-μέλη και τις προεπτικές έως προς την πολιτική και τα δημοσιοοικονομικά για το μέλλον. Όπως και τις περασμένες χρονιές έχουμε τέσσερα βασικά σημεία. Πρώτον, οι δημοσιοοικονομικές εξελίξεις ε, εστιάζοντας στην... Ξέρετε, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα και οι διερμηνείς δυσκολεύονται. Αν μπορούσατε λίγο να επιβραδύνετε. Γίνεται μια αξιολόγηση και επισκόπηση των ε, πρόσφατων δημοσιονομικών εξελίξεων εστιάζοντας την εφαρμογή ε, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου της Οικονομίας. Ε, εξετάζει ε, το πλαίσιο παρακολούθησης των δημοσιοοικονομικών, αυτό είναι το πιο τεχνικό κομμάτι της έκθεσης, ε, βλέπουμε ε, στατιστικώς πώς, πώς διαχειρίζονται τις παρεμβάσεις στα κράτη-μέλη στις αγορές. Επίσης, με μέτρηση των ε, προκυκλικών προσαρμογών των ε, δημοσίων προϋπολογισμών, εξέταση της ποιότητας των δημοσιοοικονομικών και κάτι άλλο που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ε, οι εξελίξεις στα εθνικά δημοσιοοικονομικά. Το τρίτο τμήμα που είναι το τμήμα που κανονικά βλέπουμε διάφορες αναλυτικές μελέτες στη φετινή έκθεση τονίζουμε τα διδάγματα από το παρελθόν σχετικά με την επίπτωση που έχουν τα δημοσιοοικονομικά στην κρίση του τραπεζικού τομέα. Και τέλος, όσοι ήθιστε, το τέταρτο τμήμα έχει μία επισκόπηση των ε, εξελίξεων στα δημοσιοοικονομικά στα κράτη-μέλη. Τα βασικά μηνύματα της έκθεσης, κατά τη γνώμη μας, ε, είναι ότι ε, οι δημοσιονομικές πολιτικές αποσβαίνουν τους κραδασμούς ε, της κρίσης ε, μέσα στα πλαίσια της ΟΝΕ και ε, καταπολεμούμε τα υπολείμματα της κρίσης στα δημοσιοοικονομικά. Βλέπουμε ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μας δίνει το απαιτούμενο πλαίσιο ούτως ώστε να ακολουθήσουμε αυτή την οδό παγίωσης ε, των δημοσιοοικονομικών που θα κρατήσει περισσότερο από στο παρελθόν. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις λαμβάνουν υπόψη διάφορους οικονομικούς ε, παράγοντες ε, και συγκεκριμένα το πλαίσιο των προϋπολογισμών Ένα άλλο σημαντικό μήνυμα που προκύπτει από αυτό το κεφάλαιο με τις αναλυτικές μελέτες είναι ότι ε, πρέπει να έχουμε κατά ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης ε, στα δημόσια οικονομικά είναι σημαντικές και διαρκούν πάρα πολύ. Μετά από 10 χρόνια μας δείχνουν κάποιες μελέτες μετά από μια τέτοια κρίση το επίπεδο χρέους συνεχίζει να είναι πολύ ανώτερο του επίπεδου χρέους που είχε η συγκεκριμένη χώρα πριν την κρίση. Και τα τελευταία δύο σημεία θέλω να φέρω είναι ε, ότι δεδομένης ε, ε, της μεγάλης μακράς ε, περίοδου που παγίωσε των μέσων θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να διορθώσουμε το προηγούμενο πλαίσιο που φαίνεται ότι δεν ήταν παρκώς σταθερό και κάτι άλλο σύμφωνα με την, δημόσια, την έκθεση για τα δημόσια οικονομικά Χρειάζεται καλύτερη η εποπτεία δεδομένη της τροποποιημένης δομής των δημοσιοοικονομικών λόγω της κρίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που κάνατε για τις δύο εκθέσεις και θα σταματήσω εδώ. Sven, uh, just a few minutes, if you could. Ευχαριστώ, Σφεν. Λίγα μόνο λεπτά θέλεις. Στα αγγλικά, ο κύριος Γκίγκολτ. Σημερίζομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων. που σχολίασαν την παρουσίασή μου. Πολύ λίγα είναι τα σημεία εκείνα με τα οποία διαφωνώ, έχω πρόβλημα. Το ζήτημα της κοινή εκπροσώπησης των κρατών της Ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένα στοιχείο που αναφέρεται ήδη στην έκθεση Μπερές Λάγκελ και θα το βάλω κι εγώ και χαίρομαι που το αναφέρατε. Θα πρέπει να δείξουμε όμως λίγο περισσότερο θάρρος το συζητήσαμε και αυτό όταν είχαμε και τον Επίτροπο Αλμούνια εδώ, είναι ότι η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών θα πρέπει να μας κάνει να αλλάξουμε λίγο τρόπο σκέψης, νοοτροπία. Δεν συμφωνώ απολύτως με τα όσα μας λέει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και οι κανόνες του είναι εντάξει για τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι μια διαδικασία και θα πρέπει να είναι και δεσμευτική για τις χώρες που διαφωνούν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα που ξεκινάει τη διαδικασία ελλείμματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντάξει. Αλλά υπάρχει ένας κανόνας που λέει το μισό της εκατό του ΑΕΠ θα πρέπει να αφιερώνεται στην ε, ανάκαμψη αλλά αυτό δεν είχε υπόψη του ότι μπορούσε το ε, χρέος να εκτοξευθεί στο 100%, στο 130% και ένας θεός ξέρει τι αριθμούς θα ανακαλύψουμε στη συνέχεια. Χρειάζεται λοιπόν εδώ μια ειλικρινή συζήτηση κάποια στιγμή. Και σε αυτή την ηλεκτρική και τίμια συζήτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι μηχανισμοί που θα κάνουν τις αποφάσεις πιο αποτελεσματικές και θα αλλάζουν τα όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν τα κράτη να συλλέγουν τους φόρους τους και ιδιαίτερα φόρους που ε, βοηθούν για κοινωνικές επενδύσεις και για την ανάκαμψη οικονομίας. Εδώ λοιπόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει νομίζω να είναι πιο θαραλέο από ό,τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα όσα μας λέει μέχρι τώρα και στη συζήτηση που είχαμε επαναλαμβάνει με τον Επίτροπο κύριο Αλμούνια. Ε, και χαίρομαι που θα έχουμε ειλικρινή συζήτηση και για νέες χώρες που θέλουν να ανταχθούν στην Ευρωζώνη. Τώρα δεν έχουμε χρόνο, αλλά θα ήταν χρήσιμο να μας ε, ενημερώνετε τακτικά κατά τη διάρκεια εκπόνησης τη έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά προς το παρόν. Προσβλέπω στην εργασία μαζί σας και νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα η έκθεση και για τη στρατηγική μετά τη Λισαβόνα και τη σχετική συζήτηση. Διότι θέτει κάποια, κλειδιά, κάποια ζητήματα κλειδιά που ίσως στην αρχική στρατηγική της Λισαβόνας να μην είχαν τόσο πολύ προσεχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς λέει η Πρόεδρος επόμενο θέμα, μάλλον το επόμενο χρονοδιάγραμμα για την έκθεση, σχέδιο έκθεσης 1η Δεκεμβρίου και συζήτηση στην Επιτροπή και μετά προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 8η Δεκεμβρίου. Ξέχασα να σας πω για την έκθεση του κυρίου Σχικλούνα το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι. Λοιπόν, θα σας ε, διανεμηθεί. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για το σημείο 6, επαναλαμβάνω για την ετήσια έκθεση της ε, τράπεζας, η έκθεση του κυρίου Σκυκλούνα. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 30 Νοεμβρίου 2009. Ξέχασα προηγουμένω να σα το πω. ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο σημείο για απόψε. Σα ευχαριστώ όλους εσά που παραμείνατε. Το σημείο 8 πρόθεση τη χρηστή διακυβέρνηση στο φορολογικό τομέα. Ε, θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, κύριε Ντομενίτσι. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Chair. I would speak Italian, uh, thanks to the interpreters. Θα μιλήσω την Ιταλική γλώσσα. Η έκθεση για την ε, χρηστή διακυβέρνηση στη φορολογία, στον φορολογικό τομέα, έχει άμεση σχέση με κάποιες άλλες εκθέσεις, τις οποίες έχει εξετάσει αυτή η Επιτροπή και αναφέρομαι στην έκθεση της συναδέλφου Αλβάρες, την οποία ακούσαμε προηγουμένως. Ίσως θα ήταν καλά να γίνει συζήτηση για αυτές τις δύο εκθέσεις από κοινού. Βασική αναφορά της έκθεσής μου είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28 Απριλίου 2009 για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα της φορολογίας. Προφανώς και συμμερίζομαι το πνεύμα, της κατευθύνσεις και εν μέρει το περιεχόμενο. Όπως είπαμε στην στο πρώτο τμήμα της εκθέσεως που είχε παρουσιαστεί, Υπάρχουν και άλλες αναφορές οι οποίες γίνονται στην έκθεση αυτή και έχουν, θα έλεγα, σημασία το Συμβούλιο του Μαρτίου, σαν παράδειγμα του 2008, οι αποφάσεις της ομάδας των 20 κτλ. Ο ορισμός της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα είναι στην ουσία διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών και νόμιμες μορφές ανταγωνισμού, όχι στρεβλός ανταγωνισμός δηλαδή. Αυτό έχει οδηγήσει στην συγκέντρωση της συζήτησης για την σωστή διακυβέρνηση σε δύο βασικές πλευρές, την εσωτερική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και την διεθνή από την άλλη. Για το εσωτερικό τομέα, βασικός στόχος είναι να καταργηθεί πλήρως το τραπεζικό απόρριτο, να περάσουμε στο αυτόματο στάδιο ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι κάτι το οποίο, ε, με τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να γίνεται τώρα, δεν είναι, ε, θα έλεγα, επαρκές γιατί πολλές χώρες έχουν την δυνατότητα την αυτόματη ανταλλαγή να την αλλάζουν, να την μετατρέπουν σε ανταλλαγή μετά από αίτημα άλλης χώρας. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν κάτι χρήσιμο και στα πλαίσια της καταπολέμησης ε, της, της, ε, των φορολογικών επιβαρύνσεων, της φοροδιαφυγής, των φορολογικών παραδείσων θα μας επιτρέψουν να εφαρμόσουμε με πιο σωστό τρόπο και τις προτάσεις του ΩΣΑ, περνώντας το ταχύτερο δυνατόν σε διεθνές επίπεδο στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να δει τι μπορούμε να κάνουμε σε τρεις, βασικές, σε τρεις βασικούς τομείς. Πρώτον, με τη συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με την αποταμίευση, την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία και την οδηγία που αφορά την ανάκτηση, την αρρωγή για την ανάκτηση χρεών. Συνδέονται θα έλεγα με την σωστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά τα οποία θα βρείτε στο σχέδιο εκθέσεις, έκθεσης το οποίο έχω παρουσιάσει. Θα ήθελα σύντομα τώρα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα, μια άλλη σκέψη μάλλον, όχι σε ένα άλλο θέμα. Θεωρώ ότι το κείμενο το οποίο έχει παρουσιαστεί δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένο θα έλεγα λόγω χωρικών ακριβώς περιορισμών. Θα ήθελα όμως να θέσω ορισμένες ερωτήσεις προς τους συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν στο μέλλον είτε σε τροπολογίες είτε σε συζητήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άραγε θα πρέπει να περιοριστεί στο επανέλθει σε αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα δηλαδή στα κείμενα της ομάδας των 20 της Επιτροπής και του Συμβουλίου και να λειτουργήσει και αυτό σαν ένα μικρό αλλά περιορισμένο, σημαντικό βέβαια αλλά περιορισμένο κίνητρο για την επιτάχυνση των διαδικασιών ή μήπως να γίνει χώρο συζήτησης νέων προτάσεων που να ξεπερνούν τους ορισμούς τους οποίους έχει δώσει τώρα το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα η οικονομική κρίση στην οποία ακόμα βρισκόμαστε και οι στρατηγικές εξόδου από την κρίση, οι οποίες είναι υποσυζήτηση και το είπε και ο συνάδελφος Γκίγκολτ, θέτουν σε συζήτηση τη στενή σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στις νομισματικές πολιτικές και τις φορολογικές πολιτικές, ιδιαίτερα στην περιοχή του ευρώ, στη ζώνη ευρώ. Θέτω λοιπόν τέσσερα σημεία προς εξέταση από πλευρά σας. Να συνδέσουμε καταρχάς πρώτον τη χρηστή διακυβέρνηση με το πρόβλημα μιας ευκταίας καλύτερης μορφής φορολογικού συντονισμού στο εσωτερικό της Ένωσης και μιας απαραίτητης γυτνίασης των νομοθεσιών στον τομέα των φορολογικών με όσο πιο ενοποιημένους κανόνες γίνεται. Αναφέρομαι εδώ στην ανάγκη να επανέλθουμε ε, στις, ε, στην, βάση επιβολής, στην κοινή βάση επιβολής για τις επιχειρήσεις. Καλύτερη συνεργασία λοιπόν για την φορολογία των επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν σε διακοινωτικό επίπεδο και όχι μόνο σε μία χώρα για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως το λεγόμενο transfer pricing. Δεύτερο σημείο. La governance fiscale, dei modi in cui possa essere attuata Δεύτερο θέμα είναι να δούμε πώς μπορεί να επιβληθεί μια μορφή φορολογίας στις ε, συναλλαγές ε, τις χρηματοπιστωτικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμπλέκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί τη βάση του σημείου 7 του ψηφίσματος που έχουμε εγκρίνει εμείς πριν από την κορυφή, τη συνάντηση κορυφής του Πίτσμπουργκ. Και τρίτον, να προσπαθήσουμε να δούμε μία μορφή συνεργασίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτικές έβρεσης επενδυτικών κεφαλαίων έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μην προσπαθούν να δράσουν από μόνα τους επί τη βάση αποσπασματικών κανόνων που δεν έχουν συζητηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία απλή βάση ανταγωνισμού. Και τέλος, και τελειώνω εδώ, επί τη βάση της ανάκτησης πόρων στα πλαίσια της καταπολέμησης των φορολογικών απατών, ένα τμήμα αυτών των προσόδων να έχουν σαν στόχο την τροφοδοσία του Ταμείου για την καταπολέμηση της φτώχειας και την καταπολέμηση ε, των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Είχαμε ήδη μια συνάντηση με τους σκιώδους συζητητές. Τα θέματα τα οποία θέτω προς συζήτηση ελπίζω να γίνουν αντικείμενο πραγματικής περαιτέρω συζήτησης. Έχω την αίσθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποκτήσει ένα πρωταγωνιστικό πλέον ρόλο. Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν εδώ και στρέφομαι προς τους εκπροσώπους της Γραμματείας κυρίως. Ευχαριστούμε κυρία Τζιόρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί δεν προβλέπεται η γλώσσα μου αυτή τη φορά. Άλλες φορές υπάρχει ε, παθητική διερμηνία. Μετά την παρουσίαση και τα σχόλια του εισηγητή, νομίζω ότι έχουμε όλοι μια σαφή γενική εικόνα. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη εφαρμογή των ε, εφιστάμενων κανόνων, συντονισμένες δράσεις. Αλλιώς πώς θα εξηγήσουμε στους φορολογουμένους ε, ότι ε, κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η μεγάλη απώλεια ποσών. από 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο. Επαναλαμβάνω αυτά τα τρομακτικά στοιχεία. Μεγάλο ποσοστό του ΕΕ της Ένωσης, υψηλά ποσά και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το επιτρέψουμε στο μέλλον. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι ε, από 5 έως 7 χιλιάδες δις ευρώ είναι κρυμμένα σε offshore υπεράκτης εταιρείε σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Ούτε αυτό μπορούμε να το επιτρέψουμε πλέον. Για τα εσωτερικά ζητήματα της Ένωσης μόνο 5% αντιστοιχεί σε αυτό το πρόγραμμα ανάκτησης των φόρων. Δηλαδή, το 95% χάνεται με κάποιο τρόπο ε, στις ε, ενδοκινοτικές συναλλαγές. Βάσει της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται καλά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γίνεται η επισκόπηση των ε, μέτρων που έχουν προταθεί για τα φορολογικά ζητήματα και όπου θεωρούμε ότι χρειάζεται να βελτιώσουμε τη συνεργασία. Συμφωνώ με όλες τις προτάσεις του εισηγητή και διαβουλεύτηκα με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο με διάφορους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευχαριστώ συγκεκριμένα τον κύριο Πόνη. Υπάρχουν και κάποιες καινοτόμες προτάσεις που θα ήθελα να υποβάλω και που θα μπορούσαμε να σωματώσουμε ε, να εντάξουμε στην έκθεση της Επιτροπής. Πρώτον, γιατί δεν δημιουργούμε ένα σύστημα ε, φορολογικών κινήτρων για την ανάκτηση των φόρων για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Τι εννοώ. Προς το παρόν τα κράτη-μέλη δεν έχουν κανένα κίνητρο για να προβούν στην ανάκτηση των φόρων. Γιατί δεν προσπαθούμε να μοιραστούμε τα έσοδα από αυτό Νομίζω ότι θα ήταν καλό κίνητρο για όλους και θα έδινε και μια νέα όθηση ε, στην ανάκτηση των διασυνοριακών φορολογικών οφειλών. Άλλη πρόταση που έχω να κάνω σύμφωνα με τον ΩΣΑ και το σχετικό δίκτυο για την πρόοδο που συμπιώνεται, εάν ένα κράτος συνάψει τουλάχιστον 12 συμφωνίες ε, με άλλα κράτη για την αυτόματη ανταλλαγή των δεδομένων έχει ήδη υπερβεί το όριο. Έχουμε 210 χώρες στον κόσμο, άρα γιατί μόνο με 12 χώρες δεν είναι καλός ο δείκτης, θα έπρεπε να ζητούμε περισσότερα από τα κράτη-μέλη. Τρίτη πρόταση που θα ήθελα να κάνω σχετίζεται με αυτό το transfer pricing. Έτσι κρύβονται τα κέρδη από τις επιχειρήσεις. Αυτή, αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος για, την, για να κρύβουν τα, τα χρήματα. Τι εννοώ. Όταν γίνονται οι έρευνες για υπόπτους για transfer pricing, θα ήθελα να εφαρμοστούν οι συγκρίσιμες φορολογικές μέθοδοι. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τη μόχλευση ανακλάδο και να εξετάζουμε τις μεταφορές σε θυγατρικές κατά περίπτωση για να μπορούμε να βρούμε πού έκρυψαν τα χρήματα οι επιχειρήσεις. Τέταρτη πρόταση που υποβάλλω για την ε, κατοχή μερισμάτων ή μετοχών σε offshore εταιρείε. Ε, οφείλουμε να δημοσιεύουμε τα στοιχεία σε αιτήσιε εκθέσεις ε, για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να ξέρουμε ποιος ευθύνεται. Πέμπτη πρόταση, πάλι σε σχέση με τη διαφάνεια, πρέπει να αναφέρουν οι τράπεζες τις συναλλαγές με άλλες τράπεζες φορολογικούς παραδείσους ούτω ώστε να επικρατεί η διαφάνεια σε αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω... Ευχαριστώ. Η κυρία Λούλινγκ έχει ζητήσει το λόγο. Άστρε, ζήτησε να μιλήσει το λόγο προηγουμένω στη συζήτηση αυτή. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω εκτενέστερα ως και ίδρα της ομάδας μου για το θέμα που αφορά τη διοικητική συνεργασία σε θέματα φορολογίας. Κανονικά θα έπρεπε αυτό το θέμα να συζητηθεί μετά το 8, διότι είναι το θέμα 9. Αλλά χωρίς να με ειδοποιήσετε εγκαίρως, αντιστρέψατε τη σειρά και αποφασίσατε να το συζητήσετε πολύ νωρίτερα. Μου είχαν πει στις 5, εγώ είχα έρθει 5 παρά, αλλά το έχασα. Όπως πολύ καλά είπε ο εισηγητής, όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα και συνδέονται με το ίδιο πρόβλημα. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω μερικά σχόλια που μου εμπνέει το σχέδιο έκθεση του κυρίου Ντομενισή. Ο εισηγητή, όπως και η Επιτροπή θεωρούν ότι μια καλή διακυβέρνηση ε, των φορολογικών θεμάτων περνά μέσα από τη διαφάνεια. Βέβαια κανεί δύσκολο μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Και η ίδια διαφάνεια ε, αναγκαστικά περνά μέσα από την κατάκριση του τραπεζικού απορρίτου, το οποίο εγώ αμφισβητώ. Πρώτον, στα πλαίσια της συζήτησης που κάναμε για τη φορολόγηση των καταθέσεων, είπαμε ότι η παρακράτηση στη Βυγή είναι το σύστημα που εγγυάται καλύτερα μια φορολόγηση και μάλιστα αποτελεσματική των εσόδων ε, από τόκους. Ενώ η ανταλλαγή πληροφοριών αυτή η αυτόματη πόρο απέχει από το επιθυμητό αποτέλεσμα και το προεξοφλούμενο. Ακριβώ επειδή είναι ε, βαριά η δομή και περίπλοκη η εφαρμογή της. Το ομολογεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πάντες γνωρίζουν ότι το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Αλλά οι περισσότεροι εδώ παρόντες θέλουν να καταργήσουν το σύστημα που λειτουργεί. Που είναι αυτό της παρακράτησης στην πηγή. Δεύτερον, το τελευταίο χρόνο οι προδιαγραφές του ΩΣΑ που προβλέπουν ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν ετήσεως είναι διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα. Για ποιο λόγο λοιπόν τώρα θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές και τα πρότυπα του ΩΣΑ που ε, θα υιοθετηθούν και θα εφαρμοστούν, γιατί θα πρέπει να εγκαταληφθούν και να επιλέξουμε ένα αυτόματο σύστημα που ε, έχει πολλά μενεκτήματα. Στη συνέχεια, η παρακράτηση στην πηγή εξασφαλίζει ακριβώς την ίσπραξη του ε, οφειλόμενου φόρου. Και αυτό απαντά και στις ε, εύλογες υποψίες των κρατών μελών. Και δείχνει ότι τα κράτη ε, μπορούν να διαχειριστούν χρηστά τα φορολογικά. Εγώ περιμένω να αποδείξετε το αντίθετο. Τέταρτο, ε, τελευταίο, θα ήθελα να διατρανώσω και πάλι ότι οι συστάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν είχαν μεταφραστεί στην πράξη, κανονικά στην Ευρώπη, προσεχώς, θα είχαμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε σχέση με τρίτε χώρες. Δηλαδή, οι χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαν αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ενώ οι συνδεδεμένε χώρε θα είχαν ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεω. Αυτή είναι μια στρέβλωση πάρα πολύ επιζήμια για την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι οι αρχές που υπονοεί η ε, ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αμφισβητήσιμες. Βγάζουμε συμπεράσματα ε, πριν εφαρμόσουμε ε, τα μέτρα και δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν. Τέλος, είναι γεγονός ότι συμβαίνει το εξής που θα πρέπει να μας υποψιάσει. Πρωταθλητές της ανταλλαγής πληροφοριών της αυτόματης είναι κατά κύριο λόγο οι ε, υπήκοοι της αυτής μεγαλειότητας της ε, Ελισάβετ της Δευτέρας και είναι εκείνοι που ε, εμφανίζουν τι μεγαλύτερες επιφυλάξεις να το εφαρμόσουν. Μιλάμε για οδηγία στη φορολογική συνεργασία και απέναντι σε αυτή το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρόθυμο να ανταλλάξει πληροφορίες που διαθέτει αυτό τον καιρό, δηλαδή ουσιαστικά τίποτα. Όλα αυτά λοιπόν μου φαίνονται κοροϊδία Ο εισηγητή αναφέρθηκε σε πέντε ιδέες που του είναι προσφυλή και θα ήθελα να το πω το εξής. Επειδή λέει θέλει να ενθαρρύνει την επιστροφή των κεφαλαίων. Θα ήθελα να του θυμίσω έτσι με κάθε μέτριο φροσύνη ότι έχουμε ξέρετε ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαία αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αυτό άραγε είναι συμβατό με την ιδέα αυτής της ενθάρρυνσης της επιστροφής των κεφαλαίων. Ναι, κυρία Πρόεδρε, το ξέρω ότι δεν σας αρέσουν αυτά που σας λέω, αλλά τελείωσα. Και θέλω να σας πω... Α, και κάτι άλλο για το αγαπημένο του θέμα, το φόρο Τόμπιν, μπορεί να το ξεχάσει. Άστριτ, δεν διαφωνώ μαζί σου. Έχουμε δέκα λεπτά και πολλούς ομιλητές. Και προσπαθούμε τώρα να διαπραγματευτούμε έξτρα χρόνο από τους Γερμηνείς που σχολάνε. Έχω λοιπόν στον κατάλογο Βίκυ Φόρτ και Σφεν Γκίγκολτ και Σιστόρι και Μπούλμαν και θα ήθελα να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά δεν νομίζω να χωράει. Και μετά θα επανέλθουμε και στον εισηγητή. Αυτά τα ολίγα. Uh, Ευχαριστώ. όταν άρχισα στο κοινοβούλιο πάντοτε μου έλεγαν πρόσεξε να μην μιλά κατευθείαν μετά που θα έχει πάρει το λόγο η κυρία Λούλινγκ. Δίκιο είχα. Ευχαριστώ τον εισηγητή που εργάστηκε τόσο σκληρά και συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό μαζί σας. Είναι απίστευτα σημαντικό να γίνει κάτι για τους φορολογικούς ε, παραδείσους. Συμφωνώ με την κυρία Λούλινγκ για αυτά που είπε για την αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών. Όσα η G20, το Συμβούλιο δεν ζήτησαν ακριβώς αυτό και δεν μπορεί εμείς να τα κάνουμε όλα διαφορετικά από τον υπόλοιπο κόσμο στην Ευρώπη. Δεν ε, πρέπει να περάσουμε αυτό το μήνυμα, ε, δηλαδή ας ξεκινήσουμε εμείς την αυτόματη ανταλλαγή για αφήστε τους άλλους στον υπόλοιπο κόσμο να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να συντονιστούμε. Στο 15 προτείνεται να οδεύσουμε προχωρήσουμε προς ε, μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για, την, ε, για τις εταιρείες, για φορές για τις εταιρείες. Δεν μπορεί να είναι αμφιλεγόμενη όμως αυτή η φορολογική βάση. Όλοι χρειαζόμαστε καλή διακυβέρνηση στο φορολογικό τομέα, αλλά για να μιλάμε για ενοποιημένη φορολογική βάση, ξέρετε, δεν μπορεί να μην είναι αμφιλεγόμενο το ζήτημα και για κάποια κράτη-μέλη είναι αδύνατο να το συζητήσουν. Δεν μπορεί να ορίσουν τέτοιο κοινό επίπεδο για τη φορολογία των εταιριών. Είναι κόκκινο πανί για αυτές, οπότε ε, πραγματικά δεν είναι η σωστή θέση για να υποβάλουμε αυτό το αίτημα ε, στην Ευρώπη. Στο πρότεινε εδώ μια, ένα ειδικό τέλος για τις συναλλαγές με επικράτες, με κράτη που δεν έχουν συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μιλώντας όλος ιδιαίτερος για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο D όμως αναφέρουμε ρητά ότι πρέπει να προσέξουμε με αυτή μας τη στάση, κυρίως σε σχέση με τους φτωχούς μας γείτονες. Αν δούμε ιστορικά ποιοι δεν έχουν συνεργαστεί μαζί μας, ε, λοιπόν διαπιστώνουμε ότι σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για πολύ φτωχές χώρες και οι λαοί αυτών των χωρών συχνά ε, τα μόνα κονδύλια που λαμβάνουν από εμά είναι τα εμβάσματα των συγγενών τους που ζουν και εργάζονται στη Δύση. Τώρα το να προτείνουμε εμείς επιπρόσθετο τέλος σε κάποιον προσπαθεί να στείλει αυτά τα εμβάσματα στο συγγενείς του σε μια εξαιρετικά φτωχή χώρα είναι προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε ε, το θέμα της παραγράφου 16 και ας μιλήσουμε και με τη συνείδησή μας τελικά θα βοηθήσουμε τους ε, λαούς που ζουν σε πολύ χειρότερες καταστάσεις σε σχέση με αυτή που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σβένα, σε παρακαλώ να είσαι σύντομος. Στα αγγλικά παρόλα αυτά. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισήγητη για το σχέδιο εκθεσής του, το οποίο θέτει στο κέντρο των λύσεων την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων. Πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ με ορισμένα από όσα ακούστηκα. Και συγκεκριμένα η κυρία Λούλινγκ για την παρακράτηση στην πηγή. Δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό το ιστορικό, αν δούμε τα στοιχεία από την Ελβετία και από άλλες χώρες. Τα ποσά που συλλέγονται σε καμία περίπτωση δεν είναι τα αναμενόμενα. Γνωρίζοντας τα κεφάλαια που επενδύονται εκεί. Και επίσης βλέπουμε ότι η ιδέα της αυτόματης αλλαγής πληροφοριών για φορολογικά ζητήματα η οποία για πρώτη φορά έγινε διεθνής νόμος με την οδηγία για τη φορολόγηση των καταθέσεων ε, είναι μια ιδέα που διαδίδεται τώρα και θα πρέπει να επιμείνουμε. Η Ευρώπη είναι πιο δραστήρια ε, στον τομέα αυτό για να επεκταθεί το σύστημα και σε τρίτες χώρες. Και γνωρίζουμε ε, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ότι γίνονται πολλές συζητήσεις που αφορούν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενες χώρες και ακριβώς οι αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρουν από την αδυναμία συλλογής φόρων Από πλούτο τον οποίο χειρίζονται ξένοι. Ας πούμε, στις στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει τη Εκκλησία, ε, ε, τη αναπτυξιακή βοήθεια επιμένουν σε αυτή την ανταλλαγή γιατί βοηθάει ακριβώ τι αναπτυσσόμενε χώρε και εάν είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε αυτό το μέτρο θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να επιβάλλουμε κυρώσει σε όσου δεν συμμορφώνονται. Στη συνέχεια. Στο κείμενο Συνδέεται αυτό με την ανάγκη ε, του τερματισμού του φορολογικού, του μάλλον του ε, τραπεζικού απορρίτου για φορολογικού σκοπούς. Δεν αναφέρεται ρητά, στο πνεύμα του κειμένου, ίσως δεν τονίζεται αρκετά. Και ένα επόμενο σημείο, ε, θα πρέπει να επικρίνουμε τις ασθενείς προτάσεις, τις αδύναμες προτάσεις του ΩΣΑ Συμφωνώ απολύτω με αυτό που είπαμε, ότι αν κάποιος έχει 12 διμερείς ε, συμφωνίες, ε, πολύ συχνά με άλλους φορολογικούς παραδείσους και ο σε απαλλάσσει. Ε, δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα αυτά. Θα πρέπει ανταλλαγή πληροφορώ να γίνεται αυτόματα, όχι κατόπιν αιτήσεως, γιατί έτσι δεν εξασφαλίζεται η φορολογική κυριαρχία. Υπάρχουν φόροι που δεν είναι φόροι εισοδήματο, αλλά είναι φόροι ε, περιουσία ή φόροι κληρονομία και μπορεί να συμφωνούμε να διαφωνούμε κατά πόσο είναι σκόπιμοι, αλλά κάθε χώρα θα πρέπει να είναι κυρίαρχη αν θέλει να επιβάλλει τέτοιου φόρου. Και κυρία Λούλινγκ, αυτό δεν εξασφαλίζεται από παρακράτηση στην πηγή, παρά μόνο από διαφανή και αυτόματη ανταλλαγή ενημέρωση και στοιχείων. Λοιπόν, όποιο θέλει να υπερασπιστεί τη φορολογική του κυριαρχία θα πρέπει να είναι υπέρ τη αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων. Για ένα τελευταίο. Σε αυτή την έκθεση θέλω να υπάρχει και ένα τμήμα για ένα κώδικα δεοντολογία για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Υπάρχει κώδικα, αλλά δεν εφαρμόζεται συχνά. Και υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Και προτείνω να κάνουμε έκθεση ιδέα πρωτοβουλία κάποια στιγμή στην Επιτροπή μας γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Οι προθέσεις ήταν καλές και έγινε μεγάλη βελτίωση στην αρχή, αλλά τώρα κάπου έχει αποτελματωθεί και πολλαπλασιάζεται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ο ανταγωνισμός ε, πολλών κειμένων και είναι επιζήμιος. Ε, περιμένουμε περισσότερη πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε ε, τον εισηγητή. Συμφωνούμε γενικά με το πνεύμα και θα συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε και άλλο την έκθεση. Ευχαριστώ. Έχουμε τρία λεπτά περίπου, λέει η Πρόεδρος, και έχω τον κύριο Σόριαν και τον κύριο Μπόλμαν. Μπορείτε να περιορίσετε στο ένα λεπτό ο καθένα, ε, Συγγνώμη, αλλά και ο εισηγητή θα πρέπει να απαντήσει ένα, ένα λεπτάκι. Ο κύριο Στόλογιαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλά να συγχαρώ τον εισηγητή για μια εξαιρετική δουλειά. Ιδιαίτερα για αυτά τα οποία σημειώνει στο 4. Εκεί περιγράφει την δραστηριότητα των λεγόμενων εναλλακτικών ταμείων ή επενδυτικών σχημάτων στο ευρωπαϊκό έδαφος. Θα πρέπει να συνδέεται με την επιθυμία των τρίτων χωρών να υπογράψουν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαφάνεια. Διαρωτώ βέβαια γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε οι ίδιες ρυθμίσεις δεσμευτικές να αφορούν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που εξελίσσονται στο ευρωπαϊκό έδαφος από επιχειρήσεις των οποίων η έδρα ε, βρίσκεται σε τρίτη χώρα. αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να αδειοδοτούνται μόνο εφόσον οι τρίτες χώρες υπογράφουν και αυτές με τη σειρά τους ε, τις συμφωνίες που δίδουν εχέγγυα διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών. Ο κύριος Μπούλμαν, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Λεωνάρδο Μενιτσί για την εξαιρετική του έκθεση. Θα είχα να πω δύο λόγια για την ε, ουσία, αλλά το αφήνω να τα πει εκείνο στο υπόλοιπο του, του μου. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας, σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Νομίζω ότι το σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών είναι πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σωστό να περιλαμβάνεται όχι μόνο στο δικό μου σχέδιο έκθεσης αλλά και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν μέρος στη συζήτηση και ελπίζω να συνεργαστούμε σωστά και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Πολύ ενδιαφέρουσες ε, προτάσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Λοιπόν, πάμε που δεν μπόρεσαν να χωρίς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 16 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι. Συζήτηση των τροπολογιών στις 2 Δεκεμβρίου και χαίρετε. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού αύριο το πρωί ευχαριστώ και τις μεταφράστριες για τις υπερορίες.